So, good Λοιπόν, στα αγγλικά ο Πρόεδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Άρχεται η απογευματινή μας συνεδρίαση. Θα τα πω καλύτερα τώρα ε, στα γερμανικά. Καλώς ορίσατε. Είναι ακόμα περιορισμένος ο αριθμός των παρόντων συναδέλφων, αλλά οι συνεισηγητές έχουν καταφτάσει, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Πριν ε, καλωσορίσω και δώσω τον λόγο σε πυρογνώμονες που έχουμε να ακούσουμε στο πρώτο μέρος, καλό το σύνολο της ημερήσιας διάταξης. Διαφωνεί κανείς με την ημερήσια διάταξη από τους συναδέλφους. Όχι. Ωραία, τη δέχεστε. Δεύτερον, παρατηρήσει του Προέδρου. Παρατήρηση πρώτη. Έχουμε όλοι σχεδόν τις ε, γλώσσες και σήμερα ο καθένας μπορεί να μιλάει στη μητρική του γλώσσα από τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει. Τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας και τα ντοκουμέντα, όχι εδώ. Ε, ε, όπως όλες μας συνεδριάσεις μεταδίδεται και η σημερινή στο διαδίκτυο και επίσης στις παρατηρήσεις του Προέδρου έχουμε δύο επιπλέον. Πρώτον, Την περασμένη εβδομάδα μίλησε στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργό τη Μάλτα, Ζωζέφ Μουσκάτ, ε, ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων. Γιατί έχει ε, διορίσει υπουργού και πάλι ανθρώπου ε, των οποίων τα ονόματα δημοσιεύονται σχέση με σκάνδαλα. Μας είπε ότι γίνονται τέσσερις έρευνες. Δυστυχώς, επειδή το τσέκαρα, οι τρεις δεν έχουν σχέση με τα έγγραφα του Παναμά. Οι, οι τρεις ΕΔΕ έχουν να κάνουν με υπαλλήλου ε, που ε, δεν έχουν σχέση με τον Παναμά. Δηλαδή μας παραπλάνησε. Το αποτέλεσμα ήταν οι σκληρές ε, επιθέσεις κατά του Προέδρου και άλλων μελών από διάφορα μέλη διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ζήτησε δηλαδή να αλλάξει πρόεδρος και ανακήρυξε και persona non grata. Ο συνδικαλιστής, αρχισυνδικαλιστής, σοσιαλιστής Μαλτέζος, επειδή δεν επενώ τον πρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά τον επικρίνω. Δεν κατάλαβα ε, θα αποφασίσουν πρώην συνδικαλιστές και ηγέτε των σοσιαλιστών από τη Μάλτα πώ θα οργανώσουμε εμεί τις εργασίες μας. Εγώ δεν είμαι πρόθυμος να συμφωνήσω με τίποτα άλλο αυτά. Αλλά οι ερωτήσει θα πρέπει να τεθούν εκ νέου. Και αν ο Πρωθυπουργό δεσμευτεί ε, ε, ότι θα έρθει ε, μόλις λυθούν όλα αυτά, θα τον υποδεχτούμε με χαρά ε, και με ειλικρίνεια και με δικαιοσύνη. Το λέω αυτό για να το ξέρουν συνάδελφοι που δεν έχουν μάθει τι έγινε τι τελευταίε εξέλιξει. Το δεύτερο θέμα, έχουμε στείλει δελτίο τύπου σήμερα σε σχέση, φυσικά το έχουμε συζητήσει ε, με τις πολιτικές ομάδες για την ε, πρόσβαση στα δεδομένα, τα έγραφα. Θα την έχετε πάρει την ε, ανακοίνωση τύπου, μάλιστα έχει αποσταλεί. Αυτές είναι οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Σημείο 3 έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Έξι συνεδριάσεις έχουμε, από την 6η Απριλίου μέχρι την 30η Μαΐου. Στις 19 Ιουνίου σας διαβιβάστηκαν όλα αυτά τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά? Δεις. Ωραία, εγκρίνονται λοιπόν ούτως Ερχόμαστε στο κύριο τμήμα, το πρώτο τμήμα της απογευματινής μας συνεδρίασης. Το πρωί ασχοληθήκαμε με τους whistleblowers, ε, με πέντε εμπειρογνώμονες, ενδιαφέρουσα ήταν. Ε, τώρα έχουμε τη δημόσια ακρόαση ε, ε, για το πλυντήριο της Ρωσίας. Ξεπλένει χρήματα. Έχουμε δύο επιρρογνώμονες, ο Σεμπάστιαν Φίτλερ ε, από το εγκληματολογικό της ε, Γερμανίας και τον ε, Σωματείο των Υπαλλήλων που εργάζονται στη δίωξη. Είναι στο Βερολίνο, λειτουργεί το βίντεο Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη αίθουσα γιατί προσφέρονται οι συνθήκες για τη βιντεοδιάσκεψη. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Φίντλερ, καλωσορίζω και τον Πάολο Κωνσταντζο από την ε, Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, Banca d'Italia, από ε, την Ιταλική Υπηρεσία ε, Πληροφοριών για τα Χρήματα Οικονομικά. Έχουμε προσκαλέσει περισσότερους, αλλά μόνο οι δύο ε, είναι διαθέσιμοι. Οι υπόλοιποι στην Ισπανία έχουν ε, στη Βαλένσια το Financial Action ε, Task Force συνεδρίαση και δεν μπορούν να παρευρεθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι γιατί βρίσκονται εκεί στη Βαλένθια της Ισπανίας. Επίσης, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι Λουξεμβούργο, Μάλτα, ε, ε, Ηνωμένα Βασίλειο και Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε ήδη συζητήσει με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και με το Βέλγιο και με την Γαλλία, του αντίστοιχου υπαλλήλου. Χαιρόμαστε που σήμερα έχουμε τους δύο εκπροσώπους. Γερμανία και Ιταλία, πάντα από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και δημοσιογράφους από ένα όμιλο ε, δημοσιογράφων ε, της ερευνητικής δημοσιογραφίας στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Φίτλερ και στη συνέχεια τον κύριο Κωνστάντσο. Έχετε το λόγο κύριε Φίτλερ για 10 λεπτά το πολύ από το Βερολίνο σε βίντεο διάσκεψη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη συμπερίψη της εργασίας σας. Θέλω να πω κάτι εισαγωγικά, γιατί δεν εκπροσωπώ ε, επίσημα ε, μια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είμαι αντιπρόεδρος ε, των Γερμανών εργαζομένων στην ε, Ακαδημία, την Αστυνομική και στην ε, Υπηρεσία της Δίωξης ε, ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν την, ε, τις απόψεις του κλάδου του σωματείου μας ε, και των εργαζομένων. Δεν μιλώ επίσημα υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου της, ε, των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπό την δικαλιστική μου ιδιότητα μιλώ λοιπόν. Θα ήθελα να σας πω ποια θέματα είναι για μας σημαντικά από τα σημαντικότερα είναι κυρίως φυσικά η εθνική εξέλιξη εδώ στη Γερμανία στα πλαίσια της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ε, έχει νέε αρμοδιότητε μετά από μια νέα νομοθεσία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, ένα κεντρικό νόμο για το ξέπλυμα. Στο παρελθόν αυτός ο νόμος και αυτό που ισχύει ακόμα ήταν σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή κάθε υπόνοια, ε, κάθε δήλωση ε, ήταν στο, τοπικό εγκληματολογικό τμήμα της δίωξης ε, στο καθένα από τα 16 κρατήδια και στο κεντρικό το ομοσπονδιακό ε, το ΜΠΚΑ, η Κεντρική Υπηρεσία, έχει 300 υπαλλήλους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα σε όλη τη Γερμανία και με βάση μια συζήτηση που παρακολουθήσαμε με πολύ κριτικό πνεύμα, η Γερμανική Βουλή αποφάσισε να συμφωνήσει με αύξηση του προσωπικού ε, και δημιουργία νέας μονάδας στο τελωνείο. Όχι ε, στην Ομοσπονδία και η αστυνομία δίωξης του εγκλήματος, το Bundeskriminalamt. Έχουμε επικρίσεις ε, προς τη γερμανική κυβέρνηση και δεν θέλω να τα οροποιήσω. Θέλω να πω ότι δυστυχώς κυκλοφορούν ανακρίβειες στη γερμανική βοή γιατί έγινε λόγος για ενίσχυση αύξηση του προσωπικού Δηλαδή πρόσθεσαν 20 υπαλλήλους εκεί και τους σύγκριναν με την τελική στελέχωση που θα είναι 165. Και ενώ σήμερα είναι 300 και στο μέλλον θα αυξηθούν κατά 50%. Ενώ πρόκειται για έκρηξη ε, των αναφορών ε, και των υπονοιών. 20.000 στη Γερμανία ε, ήταν πέρσι και φέτος περιμένουμε 50.000. Καταλαβαίνετε περί πρόκειται. Και κατά την άποψή μου, κάτι που πρέπει να συμπελάβουμε στη συζήτηση είναι το εξής. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μέγας λόγος για τα διάφορα μέσα και εργαλεία και τις δυνατότητες, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται αυτές οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Όλα θα είναι ωραία και καλά, αλλά θα πρέπει να δούμε να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί και που χρειάζονται. Και είναι γενική η υποστελέχωση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμαρτύρονται όλοι. Γιατί πρέπει να έχουν και κάποια προσόντα και δεξιότητες οι συνάδελφοι. Στη Γερμανία ανισχούμε πάρα πολύ και έχουμε μεγάλο ρίσκο ασφαλείας εντοπίσει τουλάχιστον για το μέλλον. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ...25 με 30% των υπόπτων ε, υποθέσεων ε, είναι διεθνής. Άρα ε, είναι αναγκαστική και η διεθνή συνεργασία. Και ε, στην Ευρώπη υπάρχει η Ευρωπόλ που χρειάζεται επιγόντως αύξηση του προσωπικού για να επεκτείνει ένα εργαλείο που υπάρχει αλλά δεν αξιοποιείται πλήρως. Τώρα, μια που έχω το λόγο, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα σημαντικότερα θέματα ε, από τη δική μας άποψη. Και εδώ ε, εκπροσωπώ ολόκληρη τη γερμανική αστυνομία αλλά και γενικότερα την ευρωπαϊκή. Στην καταπολέμηση του ξεπλήματος τι χρειαζόμαστε. Ε, κυρίως και πρώτα απ' όλα φυσικά τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι πολύτιμες, θα πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια. Βεβαίως χρειαζόμαστε ένα μητρό ε, ακινήτων για να μπορούμε να αξιολογούμε και να αναλύουμε κάθε ε, ε, αναφορά υποψία και δεν μπορούμε να έχουμε αποσπασματικές πληροφορίες και να κάνουμε τη δίωξή μας με τον παραδοσιακό τρόπο να πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις και δήμους και να ψάχνουμε στα υποθηκοφυλακεία ε, διάφορα χαρτιά, διάφορες σελίδες από κτηματολόγια. Ε, η Ισπανία έχει δείξει ότι δεν θα μπορούσαν ναι, να διώξουν ή να διερευνήσουν υποθέσεις ε, κατά Ρώσων εγκληματιών εάν δεν είχαν αυτή την κεντρική υποδομή. Λοιπόν, χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το Μητρό και οι μονάδες χρηματοοικονομικών προφοριών να έχουν τις δυνατότητες να ενισχυθούν με τρόπο βιώσιμο και αηφόρο. Αυτό είναι πραγματικά κομβικό και απαραίτητο. Κυρίως, μεταξύ άλλων, διότι οι επιτυχίες που έχουμε αυτό τον καιρό, επίσης επιτυχίες είναι αναφυσφίτητες, αλλά μιλάμε για μια τάξη μεγέθους ε, σε ποσοστά όχι της εκατό, ε, της χιλής ε, σε σχέση με τα χρήματα που ξεπλένονται και το, το, το τζίρο όλων αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό ε, θέλουμε υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα κράτη-μέλη. Αυτά εισαγωγικά ως παρατηρήσεις και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φίτλερ ένα από τα τελευταία πράγματα που είπατε ήταν το ενιαίο μητρό, το οποίο είναι αίτημα του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο για την καταπολέμηση της νομοποίησης ε, των εισόδων από παραμένες δραστηριότητες. Οι συνάδελφοι όμως θα θέσουν τις ερωτήσεις τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, καλωσορίσω και πάλι και να δώσω τον λόγο στον Παύλο Κωνστάνσο, ε, Banca d'Italia. Παρακαλώ κύριε Κωνστάνσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ ε, που με καλέσατε εδώ σήμερα. Και θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την πολύ καλή δουλειά που κάνει η Επιτροπή σας. Χαίρομαι πολύ που αποφασίσατε να επικεντρωθείτε ιδιαίτερα στις ε, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Και το λέω αυτό όχι μόνο επειδή εργάζομαι σε μια τέτοια μονάδα και επειδή βλέπω την προστιθέμενη αξία που μπορεί να δώσει η δουλειά μιας τέτοιας μονάδας και στην καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παραμονές δραστηριότητε ε, και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ζούμε σε καιρούς που πολλά αλλάζουν και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σενάρια, τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να λάβουν επαρκή υποστήριξη για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να συνεργάζονται και μεταξύ τους. Φυσικά γνωρίζω την νομοθεσία που διαπραγματεύεστε και κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε στον συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο και τις ε, τροπολογίες ε, στην οδηγία. Υπάρχουν και άλλες ε, προτάσεις που συζητώνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εργάζεται εντατικά σε διάφορα μέτωπα και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην συνεδρίαση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης αυτή την εβδομάδα. Ε, Παρ' όλα αυτά ήρθα εδώ σήμερα διότι Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας μπορεί να κάνει πολλά για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ε, αλλά και γενικά για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από ανάνομες δραστηριότητες. Όπως ε, και ο Γερμανός συνάδελφος, δεν μιλώ με την τυπική μου ιδιότητα Είμαι εκπρόσωπος ε, της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Τράπεζας της Ιταλίας. Εδώ όμως βρίσκομαι περισσότερο με την ιδιότητά μου ως μέλους ε, μιας πλατφόρμας και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία μιας προσπάθειας χαρτογράφησης ε, του φορέα αυτού σχετικά με τις δραστηριότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, και την διεθνή συνεργασία. Ε, αυτό δεν ήταν δουλειά μόνο της Ιταλικής Μονάδας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ήταν συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλία, τη Ρουμανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν. Τέσσερις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών πάντως συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Έχω ετοιμάσει μία σύντομη παρουσίαση. Θα πρέπει... Αναγκάστηκα να την απλοποιήσω αρκετά για 10 διαφάνειες πρόκειται, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να τις προβάλλουμε στην οθόνη. Okay, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ πολύ σύντομα στην προσπάθεια χαρτογράφησης που έχει, που έχει γίνει. Αρχικά η παρουσίαση αυτή ήταν πιο μεγάλη. Ελπίζω να μπορείτε να διαβάσετε τα γράμματα. Πάντως η ιδέα ήταν να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τα πρόεδρες ε, κύριε Κωνστανσό, γραπτός, ε, ε, μάλλον έχουμε μοιράσει σε χαρτί την παρουσίασή σας. Μπορούν λοιπόν όλοι οι παρευρισκόμενοι να την διαβάσουν εκ των υστέρων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και να έχει, δεδομένου ότι έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, θα ήθελα να επικεντρωθώ στη διαδικασία. Πολύ ευχαριστώ όμως θα απαντήσω σε ερωτήσεις εφόσον μπορώ, εάν ε, κάποιοι από τους παρόντες έχουν απορίες ε, σχετικά με λεπτομέρειες ε, της όλης προσπάθειας αυτής. Βλέπετε στη διαφάνεια αυτή την δομή του όλου εγχειρήματο. Επικεντρωνόμαστε στο καθεστώς την αυτονομία και την ανεξαρτησία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική τους δουλειά. Κατόπιν επικεντρωθήκαμε στις πληροφορίες που λαμβάνουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή που είναι διαθέσιμες είτε μέσω αποκαλύψεων είτε μέσω ερευνών και αναζητήσεων σε κεντρικές βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Κατόπιν η μελέτη ασχολείται με εγχώριες λειτουργίες και τι ακριβώς κάνουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών όταν ε, λένε ότι διενεργούν αναλύσει και πώς διαδίδουν, ε, πώ δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές. Ε, και κατόπιν έχουμε επικεντρωθεί στη συνεργασία μεταξύ μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, τομέα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μπορέσουν πραγματικά να δώσουν περισσότερη αξία στη συνεργασία αυτή, διότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών χρειάζονται ένα καλό δίκτυο για τη συνεργασία τους. Η εμπειρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι γενικά η συνεργασία λειτουργεί, σίγουρα όμως μπορεί και να βελτιωθεί. Υπάρχουν κάποια εμπόδια, θα πρέπει ενδεχομένως να έχουμε περισσότερη εναρμόνιση. Τέλος, ε, έχουμε εξάγει κάποια συμπεράσματα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και όσον αφορά την πιθανή μελλοντική νομοθεσία, αλλά και όσον αφορά την καλύτερη εφαρμογή της ε, και καλύτερη εφαρμογή πρακτικών από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπάρχει ομάδα εργασίας ε, όπου προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημιουργήθηκε το 2006, εδώ και πάνω από 10 χρόνια δηλαδή υπάρχει η πλατφόρμα αυτή και αναγνωρίζεται ε, με το άρθρο 51 της ε, τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων κλπ. Στόχος είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, να ε, ε, φροντίσει για τη διακυβέρνηση του δικτύου FIUNET, να βοηθήσει και να εντοπίσει διασυνοριακές αναφορές για υποπτές συναλλαγές, SDR και να διευκολύνει κοινέ αναλύσεις. Τα δύο τελευταία αυτά θέματα νομίζω ότι δείχνουν και προς τα που μπορούν να κινηθούν στο μέλλον οι εξελίξεις. Να έχουμε κεντρικό η εναρμόνιση ή συντονισμό των δραστηριοτήτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα τέλη του 2015 η πλατφόρμα υιοθέτησε το πρόγραμμα εργασίας της ε, και κάποια προγράμματα ήδη έχουν ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια της διασυνοριακή αναφορές, ε, οι προϋποθέσεις για την ε, επιτάχυνση της συγκατάθεσης για χρήση των πληροφοριών Και κατόπιν ε, έχουμε αυτή την προσπάθεια χαρτογράφησης ε, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2016. Να τονίσω κάποια πράγματα όσον αφορά τα αποτελέσματα της δουλειάς αυτής, ε, όπως επιβεβαιώθηκαν και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ τον Φεβρουάριο του 2016. μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είδαμε στην Ευρώπη. Η ε, οι υπουργοί κάλεσαν τις μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ε, πληροφοριών να επιταχύνουν τις ε, προσπάθειές τους και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενεργήσει προορατικά πάνω στο θέμα αυτό λόγω του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια αλλά και λόγω του σχεδίου δράσης του 2016 που επικεντρωνόταν σε μέτρα για ενίσχυση των δραστηριοτήτων των μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Οι εκθέσεις αυτές ε, έχουν παρουσιαστεί στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και φυσικά το Κοινοβούλιο έχει πλήρη πρόσβαση στο ε, σχετικό έγγραφο. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς αυτής θα ληφθούν υπόψη και στις τρέχουσες ε, διαπραγματεύσεις για την πέμπτη οδηγία, αλλά και κατά την εκπόνηση νέων μέτρων. και να συμπληρωθούν και με επιπλέον μέτρα, επιπλέον νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ σύντομα όσον αφορά το, το πεδίο και του στόχου. Γενικά, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών όταν συναντώνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης ε, επικεντρώνονται στον τρόπο συνεργασίας. Η δυνατότητά τους για διεθνή συνεργασία αποτελεί πτυχή των χώριων δραστηριοτήτων τους. Εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο να εξερευνήσουμε τον τρόπο με το οποίο είναι οργανωμένες σε κάθε χώρο σε κάθε χώρα οι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ε, τι δυναμικό έχουν στη διάθεσή τους ε, και τι διαδικασίε εφαρμόζουν. Διότι μόνο αν τα εξετάσουμε αυτό θα μπορέσουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών να έχουν αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του ε, και να κάνουν σωστά τη δουλειά του εντός της χώρας. Έτσι λοιπόν έχουμε ευρύ πεδίο εφαρμογής και καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών να συνεργάζονται μεταξύ τους. Επικεντρωθήκαμε και στις διαφορές ανάμεσα στις μονάδες αυτές και εξεπλάγημεν που είδαμε τι μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εξετάσαμε και την ευθυγράμμιση με διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ μας εξέπληξαν τα αποτελέσματα. Είχαμε ευρεία προσέγγιση, εξετάσαμε καταρχάς ε, το καθεστώς εντός της χώρας και την οργάνωση των μονάδων αυτών. Ε, κατόπιν ε, ανεβήκαμε επίπεδα, εξετάσαμε τη διεθνή συνεργασία και το τι μέσα έχουν στη διάθεσή τους οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, για την ε, ε, διενέργεια αναλύσεων και την διάδοση των αποτελεσμάτων. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά περαιτέρω, ανάλογα βέβαια και με τη διάθεση των Ευρωβουλευτών. Εδώ βλέπετε μία πολύ γενική σύνοψη. Έχουμε διαπιστώσει διάφορες ελλείψεις στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα εντός των διαφόρων χωρών. Φυσικά γνωρίζαμε ότι ακόμα συνεχιζόταν η εφαρμογή της οδηγίας. Δεν περιμέναμε η Εθνική Νομοθεσία ήδη να ε, ε, συμμορφώνεται με την τέταρτη οδηγία, αλλά Ε, ούτε και με την τρίτη οδηγία υπήρχε απόλυτη συμμόρφωση, για παράδειγμα κατά την ε, ενέργεια αναλύσεων ή όσον αφορά τις προϋποθέσεις ε, και τους περιορισμούς για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Βέβαια, στην Ευρώπη είμαστε αρκετά προνομιούχοι σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, διότι έχουμε μακρά παράδοση συνεργασίας. Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, ε, δεν έχουμε ρολόι στην αίθουσα, μήπως είναι δυνατόν να περάσετε στα συμπεράσματα. Ο μιλητής. Ζητώ συγγνώμη, θα ε, ε φτάσω πολύ σύντομα στα συμπεράσματά μου. Νομίζω ότι ήδη μιλάμε για συμπεράσματα διότι πρόκειται για τα αποτελέσματα της έκθεσης. Ε, μπορώ να σας ενημερώσω ότι οι αιτίε των προβλημάτων που πολύ ευχαρίστω θα αναπτύξω περαιτέρω εάν υπάρξουν σχετικές ερωτήσεις, ε, είναι και η ανεπαρκής εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα ήδη της τρίτης οδηγίας, αλλά οι ελλείψεις οφείλονται και σε έλλειψη ε, μιας ε, κατάλληλης εναρμονικής ε, προσέγγισης εναρμόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφορών διαφέρουν μεταξύ τους και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνδυάσουν το εθνικό με το διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι Έχουμε και γραπτό τα όσα μας είπατε και ε, ε, μπορούμε να κάνουμε και τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Πριν δώσω το λόγο στους συζητητές μας, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικές τάσεις και στις δύο ομιλίες. Στην τελευταία ομιλία μια προσπάθεια εναρμόνισης και δημιουργίας πλατφόρμας για να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να μάθουμε, ενώ στη Γερμανία σε σχέση με τα όσα μας είπε ο κύριος Φίτλερ, αλλάζει οργάνωση, μειώνεται το προσωπικό και αυτό δημιουργεί νέα ερωτηματικά. Αλλά θα ρωτήσουν και οι συνάδελφοι σχετικά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόφουτ. Τέσσερα λεπτά συμφωνήσαμε ε, για κάθε ερώτηση και απάντηση μαζί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Φίτλερ και τον Παύλο Κωνσταντσο. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπαν. Κύριε Φίτλερ, ζητήσατε υποστήριξη από την πλευρά μας για να υπάρχει συνεργασία με τις μονάδες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Μπορείτε να βασιστείτε βεβαίως στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ερώτησή μου. Χρειάζεται εναρμόνιση, είναι σαφές αυτό. Όσον αφορά τις ε, μονάδες συλλογής πληροφοριών για τα οικονομικά, χρειαζόμαστε νομικό πλαίσιο για ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Αλλά κύριε Κωνσταντσο, στη γραπτή σας απάντηση είπατε ότι το βασικό εμπόδιο, τα βασικά εμπόδια βασίζονται στην ανεπαρκή δυνατότητα των ξένων ομολόγων να δώσουν πληροφορίες είτε λόγω κάποιων ε, ελλείψεων ε, στο εσωτερικό ή ελλείψεων πηγών. Αυτά τα κενά, αυτές οι ελλείψεις. Μπορείτε να μας πείτε ε, τι είδου ελλείψεις εννοείτε. Έχετε παραδείγματα όπου έπρεπε να σταματήσετε τις έρευνες, τι διώξει για το ξέπλυμα χρήματο και για φοροδιαφυγή λόγω ελλείψεως ε, δυνατοτήτων δυναμικού. Ή αν υπήρχε πρόβλημα συνεργασία με τα κράτη-μέλη, αν ναι, έχετε παραδείγματα όσον αφορά τα έγγραφα του Παναμά. Ε, αναφερθήκατε στα εργαλεία. Τι εργαλεία θέλετε για να μπορέσετε να μεγιστοποιήσετε την καταπολέμηση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Στον κύριο Κωνσταντσο ρωτήσατε πρώτο και μετά τον κύριο Φίτλερ. Παρακαλώ. Thank you very much. Thanks for, for the question. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πάει ακριβώ στην καρδιά του προβλήματο. Και τα δύο αληθεύουν, κατά την άποψή μου. Έχουμε σχετικό χαμηλό επίπεδο εναρμόνιση σε κάποιου τομεί. Και γι' αυτό επιχειρησιακά αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες όταν απαιτείται από το εξωτερικό πληροφορία ίσως να μην καταφτάσει. Διότι το προσώ η αίτηση κράτος ή ομόλογός μας δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, ούτε εμείς τις κατάλληλες πληροφορίες. Είναι πολύ γενικόλογη προσέγγιση, γενική. Η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές ε, πληροφορίε και σε τραπεζικούς λογαριασμούς ε, είναι κάτι που προβλέπεται από μια οδηγία που προβλέπει εθνικά μητρώα και το Κοινοβούλιο προτείνει τροπολογίες για να διευρυνθεί το πεδίο να προσθεθούν και άλλες κεντρικές βάσεις δεδομένων που θα είναι υποχρεωτικές, υποχρεωτικό να δημιουργηθούν. Μέχρι τότε όμως Και όταν αναφέρεται έτσι γενικά ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε χρηματοστοτικέ πληροφορίε, είναι γενικόλογο ο νόμο, τότε θα υπάρχουν προβλήματα συνεργασία μεταξύ των μονάδων. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημά σα. Περιπτώσεις που έπρεπε να σταματήσουμε ανάλυση ή έρευνες λόγω ελλείψεως συνεργασίας, συνεργασίας με το εξωτερικό. Συνέβη πράγματι αυτό Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν υπήρξε καμία συνεργασία. Μονάδες για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες δεν μπορούν να απαντήσουν ή δεν έχουν την έγκριση να διαθέσουν τις πληροφορίες, να δώσουν σε, άλλες, σε άλλους φορείς πληροφορίες. Καμιά φορά είναι μερικές οι απαντήσεις. άρνηση συνεργασίας δεν θυμάμαι πρόσφατα να έχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ απαντήσει έχω λάβει. Να περιοριζόμαστε σε κάποιες πτυχέ των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Και μπορεί να είναι περιορισμένο και το πεδίο χρήσεως των πληροφοριών. Ευχαριστώ κύριε Φίντλερ. Θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα, γιατί και εσά αφορούσε η ερώτηση για τη συνεργασία. Θα προσπαθήσω ε, να σας συγκεκριμενοποιήσω αυτό που έλεγα προηγουμένως. Η εφαρμογή κάθε ευρωπαϊκής οδηγίας πάντα ε, θα υπονομεύεται και θα αποτυγχάνει εάν είναι ανεπαρκής η κρατική πόρη. Πράγμα που ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη. Για να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Αυτό το καιρό στη Γερμανία έχουμε ε, χιλιάδες ε, δηλώσεις ύποπτες που μένουν ε, στα συρτάρια και δεν την χάνουν επεξεργασίας. Και μετά σε λίγο θα ερχόμαστε σε διάφορες κοινοβουλευτικέ επιτροπές και θα εξετάζουμε για ποιο λόγο η αστυνομία, ενώ είχε περιέλθει σε γνώση της ένα ύποπτο περιστατικό, δεν το εξέτασε και δεν έδωσε συνέχεια. Μα τι πόρους έχουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή καλή είναι η κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά για να εφαρμοστεί, για να μεταφερθεί στην πράξη κάθε εργαλειοθήκη, δεν ξέρω τι άλλο, για κάθε ε, προσφυγή σε μητρό εξαρτάται από τους εργαζομένους πόσους ανθρώπινους πόρους έχουμε και με πόσα προσόντα και δεξιότητες και αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάτσεκ, συνεισηγητής και μετά εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων με πρώτο τον καθηγητή κύριο Ρωσάτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές για τις πολύ ανοιχτές παρεμβάσεις τους και τις ανησυχητικές αποκαλύψεις τους. Στην αρχή θεώρησα ότι δεξάγεται άλλη μία ακρόαση για τους πληροφοριοδότες. Είναι γνωστό ότι οι μονάδες οικονομικών πληροφοριών σε διάφορα κράτη-μέλη διαφέρουν μεταξύ τους. Έχουν προβλήματα, διαφορετικές δομές ε, έλλειψη προσωπικού, αλλά να ακούμε ξανά ότι υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνων πόρων και ειδικευμένων ανθρώπων και ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών αντιμετωπίζουν μόνο ένα χαμηλό ποσοστό των προβλημάτων, αυτό είναι πραγματικά σοβαρό. Θα είχα πολλές ερωτήσεις να απευθύνω περισσότερο στους εκπροσώπους των κρατών μελών, διότι είναι σαφές ότι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν την ίδια άποψη, κυρίως όσον αφορά το Μητρό για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, τους δικαιούς ιδιοκτήτες κλπ. Και ελπίζω αν παρακολουθούν την ακρόση δημοσιογράφοι να διαδώσουν τι ειδήσει. Ο κύριο Φίτλερ είπε ότι δεν υπάρχει μία ξεχωριστή και μοναδική μονάδα οικονομικών πληροφοριών που να διαθέτει αρκετούς α, ανθρώπινους πόρους που θα έχουν τα κατάρα προσόντα. Ποια μονάδα θεωρείτε ότι είναι στην πρώτη γραμμή που θα μπορούσε να είναι παράδειγμα. Η χώρα στην οποία εδρεύει α, και πόσο καλά εξοπλισμένη αυτή είναι η μονάδα, σαν παράδειγμα. Ευχαριστώ. Πρώτος ο κύριος Φίντλερ να απαντήσει. Παρακαλώ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να απαντήσω με τρόπο ικανοποιητικό και πλήρη, διότι αυτό σημαίνει ε, ότι ε, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο γίνονται οι αναφορές ε, για ύποπτες ε, συναλλαγές σε κάθε χώρα. Ξέρετε ότι είναι διαφορετική νομοθεσία, οι αρμοδιότητες, ποιος επεξαρτάζεται, ποια αναφορά. Το είπε και ο Ιταλός συνάδελφος, είναι πολύ ετερογενές το σύστημα στην Ευρώπη και οι αρμοδιότητες και οι δομές. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να ξεπεραστούν αν θέλουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία. Οπότε η λέξη κλειδί εδώ είναι η εναρμόνιση ε, ε, που θα σημάνει στη συνέχεια καλύτερη συνεργασία. Θα πρέπει να βρείτε κάποιες λύσεις για το τι περιμένετε εσείς από τα κράτη-μέλη, να απευθύνετε συστάσεις στα κράτη-μέλη για ποιους πόσους ανθρωπίνους πόρους θα αφιερώσουν εκεί ανεξαρτήτως ε, του συστήματος αναφοράς ε, και καταγγελίας κάθε φορά. Ρωτήστε τα κράτη-μέλη πόσες περιπτώσεις έχουν ε, στις οποίες δεν δίνουν συνέχεια. Στη Γερμανία ξέρω στοιχεία από μεμονωμένα κράτη ίδια, αλλά ευρωπαϊκά στοιχεία δεν έχω. αυτή θα μπορούσε να είναι εφετηρία για μελλοντική αντικειμενική συζήτηση. Μάλιστα κύριε Φίτλερ, αυτό μπορούμε να το ψάξουμε, να το ρωτήσουμε. Κύριος Κωνσταντσο. Um, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Φίτλερ. Το ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, ανάλογα με την κατάσταση. Αυτή η άσκηση χαρτογράφησης του ΣΥΠΗΝ δίνει κάποια στοιχεία για τους ανθρώπινους πόρους. Και ποιο είναι το δυναμικό που έχουν οι μονάδες. Από 300 μέγιστο πάμε στο ελάχιστο των 13 μελών. Μέσος όρος είναι κάπου ενδιάμεσα. Τι έχει σημασία. Ότι οι διαφορές εξαρτώνται και από διαφορές καθηκόντων και φόρτου εργασίας και εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα. Κάποιες μονάδες έχουν εποπτικά καθήκοντα πέρα από τη βασική λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Παράλληλα με τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας, όλες αυτές οι μονάδες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο όγκο αποκαλύψεων προς ανάλυση. Αυτό οφείλεται, όχι αποκλειστικά βέβαια, οφείλεται στην κατεπίγουσα ανάγκη για ανάλυση χρηματοδοτήσεως τρομοκρατών. Άρα επεξεργάζονται Περισσότερε πληροφορίε. γι' αυτό. Έχουμε και την περίπτωση των εγγράφων του Παναμά, όπου οι μονάδε εμπλέκονται περισσότερο στην, ε, σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνέ επίπεδο συνεργασίας. Να πω και ποια είναι η δική μου εθνική εμπειρία. Αλλά νομίζω ότι ισχύει και σε άλλες χώρες. Βασιζόμαστε στην πληροφορική επίση. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε χαρτιά και κατά περίπτωση εξέταση χειρονακτικά και να βασιζόμαστε μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να βασιστούμε και σε ευφυή ηλεκτρονικά εργαλεία και την σύγχρονη τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να εκμεταλλευόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη και να διερευνούμε και πιο σύγχρονε εξελίξει στο χρηματοοικονομικό τομέα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τι πολιτικέ ομάδε. Καταρχά, ο κύριο Ντάριο Ζωζάτη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισαγωγές τους. Η ερώτησή μου αφορά το θέμα που συζητήθηκε, την διασυνοριακή συνεργασία δηλαδή ανάμεσα στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πόσο συχνά λαμβάνεται αρνητική ή ανεπαρκή απάντηση από άλλη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών όταν έχετε ζητήσει πληροφορίες και ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό πέρα από το ανεπαρκές δυναμικό ή διαφορές στις ε, διαδικασίες. και μπορεί να υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή λύση σε αυτό, κάποιο πλαίσιο, ε, καλύτερη νομοθεσία, ε, εναρμονισμένη λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, ή να εισαχθούν κίνητρα ή κανόνες για τη συνεργασία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερη. Έχει να κάνει με την συλλογική χρηματοδότηση, το crowdfunding, το οποίο έχει γίνει πολύ ε, δημοφιλής τρόπος ε, συλλογής ε, χρημάτων για διάφορους στόχους. Κάποια στοιχεία δείχνουν όμως ότι το crowdfunding χρησιμοποιείται και για χρηματοδότηση όχι τόσο καινοτόμων στόχων όπως είναι η τρομοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω Είναι τομέας αυτός όπου προσπαθείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, έχετε ε, σε τακτική βάση ελέγχους, ε, ποιες είναι οι πλατφόρμες, ε, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται πραγματικά από αυτές τις καινοτόμες πρακτικές και γενικά τι παράνομες δραστηριότητες κρύβονται πίσω από αυτού του είδους ε, την ε, συγκέντρωση χρημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ερωτήσεις ακούσαμε. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει πρώτος. Κύριε Φίτλερ, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά και στις δύο ερωτήσεις, δύο ερωτήσεις άκουσα, δεν ε, γνωρίζω να υπάρχει ανάλυση στην Γερμανία. Σε ποιες περιπτώσεις έχουν ληφθεί αρνητικές απαντήσεις, από ποια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Και επίσης όσον αφορά το crowdfunding δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια ανάλυση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω ούτε σε αυτή την ερώτηση ωραία. Εάν λάβετε πληροφορίε θα τις θέλαμε πολύ στη γραπτή σας απάντηση. Παρακαλώ κύριε Κωνστανσο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, πόσε αρνητικές απαντήσεις και πόσε ανεπαρκείς απαντήσεις λαμβάνουμε. Καμία αρνητική απάντηση. Η καλή απάντηση λοιπόν είναι ότι πάντα λαμβάνουμε απάντηση στο βαθμό που είναι δυνατόν από την ε, σχετική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Λαμβάνουμε όμως πολλές ανεπαρκείς απαντήσεις από μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως η... ο πιο βασικός τύπος ανταλλαγής είναι όπου η μία μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ρωτάει την άλλη. Έχω έναν λογαριασμό στην χώρα μου, βλέπω να φτάνουν εμβάσματα από τη δική σας χώρα. Πείτε μου σας παρακαλώ από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα και από ποιον λογαριασμό προέρχονται. Και ε, δεν είναι ότι δεν υπάρχει προθυμία, αλλά συχνά δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικές και τραπεζικές πληροφορίες σε πληροφορίες ε, σχετικά με τους λογαριασμούς, ε, τις ε, συναλλαγές και από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο κράτος μέλος Α. Επίσης, το ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Κανόνες θα ήταν ο ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, περισσότερη αναρμόνιση να εναρμονιστούν οι εξουσίες ε, και ε, ε, τα καθήκοντα των μονάδων χρηματοοικονομικών προφωνιών. Όπως και ο Γερμανός συνάδελφος, ούτε και εμείς από ό,τι γνωρίζουμε, από γνωρίζω έχουμε στοιχεία και εμπειρίες από τις έρευνές μας για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων αλλά φυσικά είναι ένας τομέας που προσέχουμε ιδιαίτερα. Προσέχουμε πάντα τη συγκέντρωση πόρων, τη συγκέντρωση χρηματικών συνεισφορών, διότι για παράδειγμα κάποιες ε, κοινότητες αλλοδαπών ε, συγκεντρώνουν χρήματα, ε, είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε. Επίσης, εξετάζουμε και τα εμβάσματα. Η συγκέντρωση χρημάτων λοιπόν και τα εμβάσματα είναι δύο τομείς που εξετάζουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παουλ καν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φίτλερ, κύριε Κωνσταντσο για το χρόνο που διαθέσατε και οι παρεμβάσεις σας υπήρξαν άκρους ενδιαφέρουσες αλλά και κάπως ανησυχητικέ. Πρέπει να το πω λόγω της ελλείψεως πόρων που τονίσατε που χαρακτηρίζει τις μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πληροφοριών συγγνώμη. Πρέπει να γίνει δουλειά για τη βελτίωση της καταστάσεως. Να εστιαστώ σε ένα άλλο σημείο που αφορά την ε, υποβολή αναφορών αυτό λαμβάνει η χώρα ε, σε αμυντικό επίπεδο. Δημιουργείται θόρυβος, υπερπληροφόρηση με τα λόγια. Ή υποενημέρωση. Το εξετάζετε σοβαρά αυτό το πρόβλημα. Και ο αριθμός των αναφορών που υποβάλλεται από τις χώρες ποικίλει από χώρα σε χώρα. Η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο είχαν λίγες καταγγελίες και αναφορές. Παρόλο που είχαν αναμειχθεί σε υπεράκτιες ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στοιχήματα. Τι γίνεται με βέβαια συνεργασία μεταξύ ε, των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των φορολογικών αρχών. Σε κάποιες χώρες, ίσως σε πολλές χώρες, δεν υπάρχουν σαφείς συμφωνίες για αυτή τη συνεργασία. Άρα η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών πόρα απέχει από το να είναι ευέλτιστη. Ευχαριστώ για τη συνεργασία των φορολογικών αρχών με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ποιο θέλει να απαντήσει πρώτος. Κύριε Κωνσταντσο. Sorry. Για το πρώτο ερώτημα, για το θόρυβο και αμυντικές καταγγελίες Υπάρχει. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο, σε σημαντικό βαθμό. Και εφαρμόζονται μέτρα προς αντιμετώπιση του. Ξέρω ότι γίνεται στη χώρα μου, αλλά και οι άλλες χώρες. Στη χώρα μου παρέχουμε δείκτες στους φορείς που κάνουν καταγγελίες για να κάνουμε εκ των υστέρων εφαρμόσουμε κάποια στρατηγική. Στα πλαίσια συνεργασίας προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να μας ενημερώνουν για δραστηριότητες που έχουν κάποιο νόημα και σημασία, με τη σωστή αντίδραση, πιο γενικά. Η χρηματοδότηση των τρομοκρατών έχει επιφέρει, πώς να το πω, όχι αλλαγή μεθόδου και προσεγγίσεως, αλλά άλλαξη νοοτροπία. Χρειαζόμαστε πολλές πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι εκ των προτέρων προσέγγιση όταν υπάρχουν υπόνοιες. Χρειαζόμαστε πληροφορίες για κάποιες ανομαλίες που διαπιστώνονται, που ίσως φαίνονται αρχικά σαν αμυντική καταγγελία που δημιουργεί θόρυβο, αλλά αν χρησιμοποιηθεί σωστά η ενημέρωση αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για ε, δραστηριότητες καταπολεμήσεως χρηματοδοτήσεως τρομοκρατών Μπορεί να υπάρχει κάποια υπόνοια και αν υπάρχουν πολλές υπόνοιες δημιουργείται ένα έδος θόρυβου, αλλά μπορεί σε αχυρώνα να βρεις βελόνα αν χρησιμοποιείς σωστή προσέγγιση. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την πληροφορική για τη συλλογή πληροφοριών για την καταπολέμηση της χρηματοδοτήσεως τρομοκρατών. Δεν είναι απαραίτητα θόρυβος η αμυντική καταγγελία. Τώρα, ένα στοιχείο στρατηγικής για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι να θέσουμε κάποια όρια όσον αφορά την υποβολή καταγγελιών. Θα πρέπει οι πόνιες να ανακοινώνονται με πιο αντικειμενική υποχρέωση ενημέρωσης για τις συναλλαγές ανάλογα με το είδος των συναλλαγών και το όριο αυτών. Η συνεργασία των μονάδων χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών και των φορολογικών υπηρεσιών. Μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία λαμβάνουμε τέτοιες εκθέσεις από φορολογικές αρχές μέχρι κάποιο σημείο, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα. Για αποκαλύψεις, για διαπίστωση ξεπλήματος χρήματος από στοιχεία που απορρέουν τη φορολόγηση ή αν απορρέει από την ανάλυση των στοιχείων ότι γίνεται ξέπλήμα χρήματος. Ευχαριστώ. Κύριε Φίντλερ, θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα. Ähm, äh, Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αυτό το θέμα των καταγγελιών υπόπτων περιστατικών, αν κατάλαβα καλά, από εμάς, ε, μας ενδιαφέρει σε κεντρικό επίπεδο. Ε, ιδιαίτερα ε, οι υποψίες, καταγγελίες σε τομείς που δεν έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Στην Γερμανία παραμένει αυτό αρμοδιότητα των κρατηδίων και το 2012 η Άνω Βουλή ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να γίνει ομοσπονδιακή ε, αρμόδιότητα. Είναι και δική μας θέση. 16 είναι τα ομόσπονδα κρατήδια στη Γερμανία, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, άρα η εποπτεία δεν είναι καλή γιατί είναι και αυτά υποστελεχωμένα. Πάνω από 90% των καταγγελιών προέρχονται από τα χρηματοοικονομικά και τα μη χρηματοοικονομικά σχεδόν δεν έχουμε καμία ε, καταγγελία. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε επίβλεψη, δεν έχουμε ε, ευαισθητοποίηση των εθνών των εμπόρων, ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες ε, αναλύσεις ε, δεν υπάρχει ε, ευαισθησία για αυτό το θέμα και στη Γερμανία πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία για τους άλλους κλάδους, όχι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το άλλο αφορά τη συνεργασία των φορολογικών αρχών και πάλι θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση στη Γερμανία. Υπάρχει ακόμα αποκεντρωμένο μοντέλο που ισχύει, δηλαδή η αστυνομία δίωξη του εγκλήματος συνεργάζεται με το τελωνίο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατηδίων σηκώνει βελτίωση το θέμα αυτό, αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται από το παρελθόν. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις για τη μελλοντική δομή των μελλοντικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Άρα περισσότερα ερωτηματικά έχουμε και εμείς για το μέλλον παρά απαντήσεις να δώσουμε. Και είναι και τμήμα της κριτικής. Ευχαριστώ κύριε Φίτλερ. Όσοι γνωρίζουν το ομοσπονδιακό σύστημα στη Γερμανία ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να συνεργάζονται 16 ομόσπονδα κρατήδια. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία που είναι ομοσπονδιακή χώρα επίσης. Ο καθηγητής ε, κύριος ε, Λούκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία σειρά ερωτήσεων που θα ήθελα να θέσω. Καταρχάς ε, και απευθύνομαι και στους δύο μιλητές, θα ήθελα να γνωρίζω τη θέση σας σχετικά με την πιθανή πολιτική επιρροή των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Από τη συνεργασία σας με άλλες μονάδες σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζετε συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις όπου ε, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα πολιτικής επιρροής εδώ ή όπου να βλέπετε τη μονάδα να λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολιτική επιρροή. Αυτό με ενδιαφέρει, διότι κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ε, βρίσκονται υπό υποψία να είναι ασφαλείς λιμένες για τέτοιες δραστηριότητες. Εάν μπορείτε να μας πείτε λοιπόν ότι ειδικά σε κάποιες χώρες οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών μπορούν να βρεθούν υπό ε, πολιτική πίεση, αυτό θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας. Δεύτερη ερώτηση. Με ενδιαφέρει η εσωτερική οργάνωση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Στη δική σας ή σε άλλες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών γίνεται αξιολόγηση της δουλειάς αξιολόγηση των προβλημάτων και των επιτυχιών. Υπάρχει κάποια έκθεση που δείχνει εκρεμείς ε, υποθέσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Φίτλερ για τη Γερμανία. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κολλήσει, ε, που σχετίζονται και με μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπάρχουν στοιχεία σχετικά με ε, τα χρήματα που έχουν ανακτηθεί είτε στη δική σα είτε σε άλλη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών υπάρχει τέτοια έκθεση. Εάν όχι, τι σα εμποδίζει να εκπονήσετε τέτοια έκθεση. Και ε, σημαντικό ίσως θα ήταν να αυξήσουμε την πολιτική πίεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετικά ε, τελικά έχει περιορισμένες εξουσίες. Κάποια πράγματα αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά Επειδή πολλές ε, από αυτές τις υποθέσεις έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και ε, συχνά κολλάνε, ίσως επειδή δεν είναι ικανοποιητική η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ίσως θα ήταν ε, χρήσιμο εμείς να ζητήσουμε την δημοσίευση τέτοιων εκθέσεων. Μία τελευταία παρατήρηση. Σημείωσα διάφορα ε, θέματα στα οποία είπατε ότι θα πρέπει να συνεργάζονται οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ε, να υπάρχουν να εναρμονιστούν ε, οι αρμοδιότητες ενέργειας, τα, τα κεντρικά μητρώα και οι πληροφορίες να μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα ήταν σημαντικά για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ε, μήπως υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να λύσουμε με νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ποιος θα ξεκινήσει. Κύριε Φίτλερ. Ναι, ευχαρίστω κύριε Πρόεδρε. Θα δηλώσω εθελοντή για να απαντήσω πρώτο. Ε, θα προσπαθήσω ε, στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να σα ε, απαντήσω. Πολιτική πίεση. σε περιορισμένο βαθμό μπορώ να μιλήσω μόνο. όσον αφορά την Γερμανία, και όσον αφορά την κατάσταση μέχρι τώρα ε, και την, ε, τις αρμοδιότητες μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει πολιτική επιρροή. Ε, θέλετε να το πω έτσι ότι ε, η πολιτική επιρροή ασκείται στο ότι ουσιαστικά περικόπτονται οι πόροι μας και το δυναμικό μας. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική πίεση. Ε, χειρότερη πολιτική θα μπορούσα, ε, χειρότερη πολιτική πίεση δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Όσον αφορά άλλες χώρες ε, δεν μπορώ να σας πω. Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση και την υποβολή εκθέσεων. Κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Στην Γερμανία τα βασικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται σε δύο εκθέσεις και οι δύο δημοσιεύονται από την Ομοσπονδιακή Συνομία, το Bundeskriminalamt. Και αναφέρεται η αξιολόγηση ε, των ύποπτων ε, ε, υποθέσεων με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εγώ ήδη σας έδωσα πληροφορίες. Το 90% των υποθέσεων έχουν να κάνουν με το χρηματοοικονομικό τομέα και πλέον έχουμε μια άλλη έκθεση που δείχνει πόσο επιτυχής ή πόσο λίγες επιτυχίες έχουμε Υπάρχει το πρόβλημα ότι έχουμε επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και είναι κάτι για το οποίο ε, παραπονόμαστε εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό κοιτάμε πάντα την Ιταλία, διότι οι Ιταλοί συνάδελφοι έχουν ε, καλά μέσα στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά. Νομίζω ότι η τελευταία ερώτηση ήταν ε, αν χρειάζεται τίποτα επιπλέον. Ε, όσον αφορά τις προτεραιότητες ε, θα έλεγα μετά από το ανθρώπινο δυναμικό και τα κεντρικά μητρώα, ε, τις δυνατότητες έρευνες, αυτά είναι τα βασικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην εισαγωγή σας ε, αναφερθήκατε και στην πρόσβαση σε μητρώα ακινήτων. Μετά από τους επένους που ακούσαμε για την ε, Ιταλική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ε, νομίζω ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε και σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα για τα διάφορα σημεία που εφήγησαν. Για την ανεξαρτησία έναντι πολιτικής επιρροής. Να τονίσω καταρχάς ότι στην περίπτωσή μου Είμαστε εντό τη κεντρική τράπεζα. Έχουμε διπλή στιβάδα, αν θέλετε, ανεξαρτησία από την πολιτική εξουσία. Διότι είναι εξάρτητη η κεντρική τράπεζα πρώτα απ' όλα, διότι εμεί είμαστε εξάρτητοι εντό τη κεντρική τράπεζα. Άρα είμαστε πολύ καλά ε, προστατευμένοι. Έχω την πεποίθηση ότι λίγο πολύ η ίδια κατάσταση ισχύει και για άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσης. Δεν γνωρίζω για υποθέσει πολιτική επιρροή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω για θέματα σοβαρή πολιτική επιρροή σε άλλε χώρε μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών καμιά φορά χρησιμοποιούνται για πολιτικέ διαμάχε. Χρησιμοποιεί τα στοιχεία των μονάδων αυτών η κυβέρνηση για τα επίτευξη τακτικών πολιτικών στόχων για να υπονομεύσει το κύρος αντιπάλων καμιά φορά. Και χρησιμοποιεί και ξένες πληροφορίες για να το κάνει αυτό. Αυτό αποτελεί απειλή όταν συμβαίνει σε μια χώρα. Αυτό που συμβαίνει καμιά φορά είναι κάτι διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικητική επιρροή, όχι πολιτική. Οι μονάδες δημιουργούνται εντός μιας μεγάλης οργάνωσης, μεγάλου οργανισμού, δεν επηρεάζονται από πολιτικούς, αλλά μπορεί να επηρεάζονται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της, ε, του οργανισμού στον οποίο ανήκουν και να αποφασίζουν για προπολογισμό, για πόρους, για προτεραιότητες. Υπάρχει μια επιρροή που καμιά φορά φαίνεται και από τη συλλογή των στοιχείων αυτή τη χαρτογράφηση που κάναμε. Είναι διαφορετικού είδους πρόβλημα, αλλά σοβαρό για την αξιολόγηση του έργου. Η αδίποτε διοίκηση, οσδήποτε οργανισμός έχει τρόπους να δοκιμάσει να ελέγξει το έργο που παράγει. Εμείς στην Ιταλία το μεταφράζουμε αυτό στην έννοια της λογοδοσίας. προσπαθούμε να λογοδοτούμε προς τα έξω. Έξω τι εννοώ. Αυτό εξαρτάται από τις εθνικές διευθετήσεις αυτό. Αλλά στην περίπτωσή μας λογοδοτούμε στο κοινό εν γέννη, δημοσιεύουμε στοιχεία, στατιστικά στοιχεία, που αυτά προσπαθούν να αντικατοπτρίσουν το φόρτο εργασίας και τα αποτελέσματα του έργου μας. Επίσης είμαστε υπόλογοι και στο Κοινοβούλιο, λογοδοτούμε στο Κοινοβούλιο, διότι διακυβεύονται χρήματα και το δημόσιο συμφέρον και θέλουμε να δείξουμε ότι προστατεύουμε αυτά τα συμφέροντα. Άρα υποβάλλουμε εκθέσεις και στο Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία. Δύο προβλήματα να τονίσω και ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, οι μονάδε χρηματοοικονομικών δεδομένων υφίστανται διότι κάποιο πρέπει να κάνει την ανάλυση. Και αυτό είναι διαφορετικό από την έρευνα και καμιά φορά είναι θολή αυτή η διάκριση. Είναι κρισίμου σημασία. Αν θέλουμε να δώσουν Έρευνε με προστιθέμενη αξία αυτέ οι, χρηματοοικονομικές, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να γίνεται αυτή η διάκριση. Αλλιώ συγχαίρεται η εικόνα και μειώνεται η αποτελεσματικότητα τη ε, μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Και τώρα πώ χρησιμοποιούμε τι πληροφορίε που ανταλλάσσονται μεταξύ μονάδων. Λαμβάνουμε απαντήσει στα αιτήματά μα, αλλά πολύ συχνά αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνες ή για δίωξη διότι δεν έχουμε τη συνένεση τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχει πληροφορίε. Δεν έχει την εντολή να κάνει τέτοιο. Άρα ο περιορισμό χρήσεω των πληροφοριών που ανταλλάσσονται ε, είναι ένα εμπόδιο όσον αφορά την διεθνή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, ερωτήσεις και απαντήσεις ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε ε, και νομίζω θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Μπορεί ένας από τους βασικούς λόγους για την καλή οργάνωση της μονάδας στην Ιταλία να είναι η μαφία. Ε, η Γκουε, παρακαλώ, Μαρκάτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Κωνσταντζο. Έγιναν μελέτες για την Επιτροπή μας και σχολιάζουν τη σχέση μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των μονάδων επιβολής του νόμου. Και οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι ενταγμένες στις αστυνομικές υπηρεσίες έχουν καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Εσείς αναφερθήκατε στην αυτονομία ε, των μονάδων. Πέρα του να εξασφαλίζουμε ότι έχουν νομική αυτονομία και εξουσία οι μονάδες αυτές, Πιστεύετε ότι οι μονάδες αυτές που δεν είναι ενσωματωμένες στις μονάδες επιβολής του νόμου μπορούν να πετύχουν καλύτερα επίπεδα αυτονομίας. Ή θεωρείτε το μοντέλο ύπαρξής τους δεν επηρεάζει αυτή την κατάσταση. Μια ερώτηση για όλους. Οι δείκτες κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατών διαφέρουν σημαντικά και είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να προληφθεί η χρηματοδότηση τρομοκρατών, διότι ίσως να χρησιμοποιούνται νόμιμοι πόροι σε μικρά ποσά και μετά να επιτυχάνονται εγκληματικοί σκοποί. Μπορείτε να περιγράψετε πώς λειτουργεί το σύστημα στις χώρες σας. Μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών ε, και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του φαινομένου για να είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα ο Κωνστανσό και αν θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Φίτλερ με χαρά να το κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Λοιπόν, η ανεξαρτησία των μονάδων. Κάναμε έρευνα και τι έδειξε. Ότι το μοντέλο λειτουργίας των μονάδων επηρεάζει την ανεξαρτησία δεν είναι επιλογή αυτή του μοντέλου, αυτή καθ' αυτή. Δεν ισχύει ότι οι αστυνομικές μονάδες χρωματοοικονομικών πληροφοριών είναι λιγότερο εξάρτητες από άλλες μονάδες που δεν είναι στην αστυνομία. Έχουμε στοιχεία όμως, σύμφωνα στις πληροφορίε που έχουμε συλλέξει, που δείχνει ότι οι αστυνομικές χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ενσωματωμένες περισσότερο στις αστυνομικές αρχές. Καμιά φορά σε γραφεία της αστυνομίας και ίσως να είναι λιγότερο ανεξάρτητες εν συγκρίση με άλλες χρηματο, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι ανεξάρτητες, ανεξάρτητοι φορείς. Είναι διότι είναι πολύ βαθιά ενσωματωμένες οι μονάδες στις νομικές αρχές που τις κάνει λιγότερο ανεξάρτητες. Και άλλους παράγων. και αυτό είναι ο κίνδυνος αστυνομικών ε, χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μπορεί να αναμίξουν ανάλυση και έρευνα. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Χρησιμοποιούν στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές για να ξεκινήσουν πραγματικές έρευνες, χωρίς να διαχωρίζουν την ε, ε, οικονομική ανάλυση από τις έρευνες. Τώρα για τους δείκτες κινδύνου ε, όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματο στην με τη χρηματοδότηση τρομοκρατών. Είναι ένα παρόν πρόβλημα, πολύ σχετικό αυτό που θέσατε. Πρέπει να δοθούν πολλέ πληροφορίε στου αρμόδιου φορεί για αυτού του σκοπού. Το ξέπλυμα χρήματο παραδοσιακά είναι κάτι πιο εύκολο, διότι έχουμε ίσω περισσότερη εμπειρία. Η χρηματοδότηση των τρομοκρατών είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Όπω είπατε, ε, τα ποσά είναι πολύ πιο μικρά δεν υπάρχουν, εντοπίζονται εύκολα ανομαλίες. Είναι κανονικές συναλλαγές αυτές που έχουν προορισμό τους τρομοκράτες. Μέσω αντικειμενικής αναλύσεων δεν μπορούν να εντοπιστούν. Ε, μπαίνουν μέσα κάποια υποκειμενικά στοιχεία και αυτά σχετίζονται με πολύ ευαίσθητα στοιχεία που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Είναι ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το επεξεργαστούμε και σε διεθνές επίπεδο, ενώνοντας τις δυνάμεις μας και συλλέγοντας Πληροφορίε των μυστικών υπηρεσιών και προσπαθούμε να τι ανταλλάσσουμε τόσο ώστε να έχουμε και την κατάλληλη επαφή και τροφοδότηση. Κύριε Φίτλερ, έχετε να προσθέσετε τίποτα. Μου δώσατε το λόγο. Ναι. Δεν είστε υποχρεωμένο, αλλά αν θέλετε παρακαλώ. Πολύ σύντομη συμπλήρωση για να συμφωνήσω με τον προαλήσαντα. Καταρχήν, για την τρομοκρατία, ε, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε μια πιο πυκνή συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να διασταυρώνουμε κριτήρια πρόσωπο παγή με ε, κριτήρια σχετικά με τις συναλλαγές, τα οποία θα πρέπει συνεχώς να επικυροποιούνται και να ενημερώνονται. Και το στοιχείο της ανεξαρτησίας μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τις μονάδες χρηματοοικονομικών προφορών Δεν θέλω να επανέλθω στη Μάλτα, αλλά εκεί τέλειωσε μια έρευνα η μονάδα η οποία δεν διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, διότι δεν ήταν δεδομένη ανεξαρτησία. Άλλο θέμα αυτό όμως, καμία σχέση. Θα δώσω το λόγο στο Σβεν Κίγκολτ από πλευρά των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω υπόψη μου τουλάχιστον τρεις εκθέσεις ε, της μονάδας χρηματοοικονομικών Προφορών στη Μάλτα, στις οποίες δεν δόθηκε συνέχεια. Ε, αν μας ακούνε, να μας τα στείλουν ή να σας τα δώσω εγώ τα στοιχεία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντσου. Διαβάσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας. Πιστεύω ότι το έργο σας είναι πολύτιμο. Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, με λεπτομέρειες, όσο πιο ακριβής γίνεται, μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε αυτά που είπατε στη γραπτή απάντησή σας. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Ποιες παραβάσεις, ποιες παραβιάσεις ή ατελείς εφαρμογές της οδηγίας, της τρίτης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος διαπιστώσατε σε ποια χώρα. Λέτε ότι είναι ατελείς η εφαρμογή και δεν είπατε ποια είναι τα κράτη-μέλη, ποιε είναι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δεν συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την οδηγία. Στη σελία στη σελίδα με παριθμό 37, λατινικός αριθμός, ζητάτε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή τέτοια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Γιατί πιστεύετε ότι μια τέτοια μονάδα ευρωπαϊκή ε, χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση ήταν προς τον κύριο Κωνσταντσο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παραβιάσεις της ε, τρίτης οδηγίας. Δεν θέλω να κατανομάσω χώρε, δεν τι έχω μπροστά μου. Εργαστήκαμε βάσει ε, πληροφοριών που όμως δεν κατονομάζονται συγκεκριμένε παραβάσεις στην ε, έκθεση. Μόνο τα στοιχεία στατιστικά παρουσιάζονται. Παραδεχόμαστε όπου κάπου η εθνική εφαρμογή ή πρακτικές δεν ευθυγραμμίζονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Παράδειγμα, όταν μια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοστατικές πληροφορίες. Τι εννοώ με αυτό. Απλές πληροφορίες που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει σε εκείνους που συνέλεξαν τις πληροφορίες ότι ε, παραβιάζεται η τρίτη οδηγία, ίσως και η δεύτερη μάλιστα. Και σίγουρα οι σχετικές συστάσεις των αρμοδίων αρχών Υπάρχουν και υποθέσεις και προβλήματα όσον αφορά τη σύμφωνη γνώμη που πρέπει να χορηγείται για τη χρήση των πληροφοριών. Προβλέπει, η τρίτη οδηγία προβλέπει γενικό καθήκον των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών να επιτρέψουν να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που χορηγούν για περαιτέρω έρευνες. Εκτός για κάποιες εξαιρέσεις. Στην πράξη καμιά φορά οι εξαιρέσεις είναι περισσότερες από τον κανόνα πολύ συχνά αρνούνται τη σύμφωνη γνώμη, την έγκριση, από ότι να εγκρίνουν τη χρήση των πληροφοριών. Η έκθεση δείχνει ότι σε κάποιους τομείς δεν εφαρμόζεται σωστά η τέτοια οδηγία. Ίσως να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Αν έχω χρόνο μπορώ να προχωρήσω. Προσπαθώ να εστιαστώ επί των πιο σημαντικών πτυχών Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση του κυρίου Γκίγκολτ. Πολύ συγκεκριμένη. Αυτό τον κατάλογο μπορείτε να μας το στείλετε, ακόμα και αν δεν είστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κατονομάσετε χώρες. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, μην το κάνετε. Παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε γραπτός. Ε, τομείς που έχετε προβλήματα με μια τρίτη χώρα. Κοιτάξτε, με τα χαράς να δώσω στην Επιτροπή έναν απλό κατάλογο των πορισμάτων μας που αναφέρονται στην έκθεση. Λοιπόν, για την ε, η μονάδα χρηματοοικονομικών ε, πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ευρωπαϊκή μονάδα. Έχουμε σε μια, μια παράγραφο που λέει ότι μια τέτοια μονάδα θέλει να απαντήσει σε αυτά τα προβλήματα. Επιτρέψτε μου να το αναλύσω αυτό περαιτέρω. Να πω ότι εκ των υστέρων μπορεί να πει κανείς ότι χρειάζεται και κάποια άλλη ανάλυση. Διαφέρουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών από χώρα σε χώρα. Δύσκολο να έχει κανείς τέτοια ποικιλομορφία. Δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματική λύση τώρα. Ίσως χρειάζεται ε, καλύτερη εναρμόνιση και συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Του, του λεχθέντων συντονισμός και διευκόλυνση συνεργασίας είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φίτλερ, θέλετε να απαντήσετε. Η ερώτηση απευθυνόταν μόνο στον συνάδελφο Σα Θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Να πω μόνο ότι ε, διαβεβάζουμε στην Europol ε, τις αναφορές και τις καταγγελίες σε μια βάση δεδομένων ε, και κάνει τις διώξεις και τις έρευνες. Βεβαίως, εξαρτάται και η Europol από τις αρμόδιες εθνικές διεκτικές αρχές για να τους τα διαβιβάζουν. Μάλιστα, τελείωσαν οι πολιτικές ομάδες. Έχω ε, κάποιον από το ΚΑΤΣΙΑΕ, συγκεκριμένα την αντιπρόεδρό μας, Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ. Μας λέτε λοιπόν ότι 90% των εκθέσεων προέρχονται από το χρηματοδοτικό τομέα. Άλλοι φορείς όπως ε, ε, οι νομικοί ε, και οι μεσίτες δεν είναι τόσο υποχρεωμένοι. Κανείς δεν τους υποχρεώνει να δώσουν πληροφορίες. Κύριε Κωνσταντζο, τι γίνεται με το νέο πρόγραμμα το επενδυτικό, για τους επενδυτές που εφαρμόζεται στην Ιταλία. Ε, είναι μια χρυσή βίζα που δίνεται, αν θέλετε, που θα μπορούσε να τροφοδοτεί τελικά το ξέπλυμα χρήματος. Ποιο είναι ο ρόλο των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να ελέγχουν μεταφορές υπεράκτιε σε υπεράκτιου λογαριασμού. Πρέπει να κοινοποιούνται αυτέ οι κινήσει από χρηματοδοτικούς ε, ε, χρηματοστατικά ιδρύματα και τράπεζες και να κοινοποιούνται αυτές οι κινήσεις φορολογικές αρχές. Όχι στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών κάνετε ένα τέτοιο έλεγχο για τη μεταφορά πόρων προς τις υπεράκτιες αυτές τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία ερώτηση αν σκεφτείτε και τίποτα άλλο, θα υπάρξει και τελικό γύρος. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντζο. Uh, yes, thank you. On uh, the uh, reporting... Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τις αναφορές που λαμβάνουμε από μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μπορώ να σας πω από την πλευρά της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ότι αυξάνεται η συνεργασία από πλευράς του μη χρηματοοικονομικού τομέα. Λαμβάνουμε περισσότερες αναφορές από, για παράδειγμα, συμβολεογράφους, λογιστές, αλλά και από μη ε, χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Ένα στοιχείο που βοηθάει είναι ο ρόλος που παίζει η αυτορύθμιση, <coughs> ε, που διευκολύνει τους ε, διάφορους επαγγελματίες να αναφέρουν περιστατικά διασφαλίζοντας ε, το απόρριτο. Επίσης ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο. Όσον αφορά τα τις μεταφορές και κεφαλαίων ε, από υπεράκτιες εταιρείε. Αυτό είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς κινδύνου που παρακολουθούμε συνέχεια. Εξετάζουμε λοιπόν ε, τις δικές μας πηγές ε, αλλά και στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Υπάρχουν διάφορα καθεστώτα για τις υπεράκτιες ε, εταιρείε, υπάρχουν διάφορες χώρες, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία και γι' αυτό απαιτείται διεθνής προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο να μπορεί να λύσει ούτε μία μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών μόνη της, ούτε μία χώρα μόνη τους. Ε, πρόεδρος, όσον αφορά την ε, αυτορύθμιση των ε, διαφόρων επαγγελματιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση σήμερα όπου ε, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αναφέρουν υποψίες. Και αυτό μαζί με τις άλλες ε, κυρώσεις θα είναι αποτελεσματικό μέσο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φίτλερ. Ναι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ε, μ' αρέσει να διαφωνώ, αλλά η Γερμανία δεν είναι πολύ αισιόδοξη στο θέμα αυτό. Ε, μόνο Ε, οι φορείς αυτορύθμισης μάλλον από τους τομείς ε, αυτορύθμισης, από τους δικηγόρους, από τους ε, λογιστές κτλ. λαμβάνουμε πολύ μικρό ποσοστό αναφορών με παροχή συμβουλών, με ευαισθητοποίηση θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερες αναφορές, να τους ενημερώσουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με αυτό. Μόνο έτσι θα το καταφέρουμε και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχο καθεστώς ελέγχων. ώστε κάποιο που έχει λάβει τέτοιε πληροφορίε να είναι απολύτως υποχρεωμένος να τι υποβάλει. Ε, κύριε φίλε, σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, διαφωνείτε. Συμφωνώ πολύ με τη θέση σα. Από ό,τι είδα, η αυτορύθμιση είναι ανεπαρκή σε κάποιου τομεί στην ε, διαδικασία συναπόφασης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Και αν έχετε σχετικές προτάσεις, ε, πολύ ευχαριστώ θα τις λάβουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σημερινούς ομιλητές μας ε, του πρώτου πάνελ. Ακούσαμε διάφορα χρήσιμα πράγματα για την συνέχεια των εργασιών μας. Κύριε Φίτλερ, ε, πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας σήμερα. Μας μιλήσατε για αύξηση του προσωπικού και λόγω της νομοθεσίας για τη μάφια βλέπουμε ότι και η Ιταλία έχει εξαιρετική νομοθεσία. Απομένουν βέβαια πολλά να γίνουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ε, μας υποσχεθήκατε γραπτές απαντήσεις και ε, πρόσθετες πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να μας τις στείλετε. Θα ήθελα να κλείσω τώρα το πρώτο τμήμα της ε, σημερινής μας ακρόασης ε, και τρία λεπτά διάλειμμα θα κάνουμε και κατόπιν θα προεδρεύσει η Άννα Ο πρόεδρος ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Um, let's start now the second session. Πάρτε τις θέσεις σας παρακαλώ, καθίστε. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Έχουμε την περίπτωση του ρωσικού πλυντηρίου. Mm-hmm. Οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ είναι ο Πολ Κρίστιαν Ραντό από το ερευνητικό φορέα για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά και το σχετικό πρόγραμμα, ο κύριος Βίστος Μπούρκανς από τη Λετωνία και για το ξέπλυμα είναι για το ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες. Έχουμε βιντεοδιάσκεψη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρκαντς που είστε διαθέσιμος. Ας ακούσουμε λοιπόν Κύριε Ραντού, να επαναλάβω τη μεθοδολογία. Κάθε ομιλητής έχει το πολύ 10 λεπτά στη διάθεσή του. Να κάνει τις αρχικές του παρατηρήσεις. Μετά την παρουσίαση των ομιλητών θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Θα υποβληθούν ερωτήσεις ανά πεντάλεπτα. Η ερώτηση ένα λεπτό και χρόνος για απάντηση. Και κύριε Ράντου έχετε το λόγο χωρίς να καθυστερούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εκπροσωπώ το όλο πρόγραμμα για τον εντοπισμό του ξεπλήματο χρήματο και υποβολή αναφορών. Είμαστε το μεγαλύτερο φορέα στον κόσμο για αυτό το θέμα και τι κάνουμε. Ακολουθούμε το χρήμα. Το 2010 μαζί με συναδέλφους είδαμε κάτι. Ότι συνεχώς ερευνούσαμε το ίδιο πράγμα. Ήταν το ίδιο το έγκλημα και ξέπλυμα χρήματος υψηλού επίπεδου από τις διάφορες συμμορίες των ναρκωτικών στον κόσμο, Μεξικό κλπ. Το 2010 αποφασίσαμε να ερευνήσουμε την υποδομή που επιτρέπει το ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα. Και είδαμε ότι υπήρχε μια νεοζηλανδική εταιρεία και είχε λογαριασμό σε μια τράπεζα στην Λετωνία. Περίπου 680 εκατομμύρια δολάρια ε, κινούνται σε αυτό το λογαριασμό συναλλαγές. Και δεν είναι κατά χρήματα σε ένα δικαιούχο, αλλά σε πολλές εγκληματικές ομάδες ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, χρήματα του Μαγνίτσκι κλπ. Διάφορε ομάδες, διάφορες συμμορίε ε, πέρναγαν τα χρήματά τους από εκεί. Πολύ ενδιαφέρον. Υπήρχε μια πλατφόρμα, έτοιμη πλατφόρμα. Αυτή επέτρεπε ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα, σε πολύ χαμηλό κόστος, εν συγκρίση με τις παραδοσιακέ μεθόδου ξέπλυματος χρήματος. Αυτοί που ξέπλαιναν τα χρήματα έφτιαχναν την, την πλατφόρμα, βάζαν τράπεζε, έδιναν στου πελάτε υπεράκτιε εταιρείε με τραπεζικού λογαριασμού στι τράπεζε που ήλεγχαν και εξέδιδαν και εγχειρίδια απάτη, όπω αποκαλούνται. Έδινε η τράπεζα μια έτοιμη υπηρεσία για το ξέπλυμα χρήματο και το εγχειρίδιο συμπεριλάμβανε πληροφορίε διάφορε. Μη, να, να, λένε, μη στέλνετε ε, στον κυλούς αριθμούς ένα εκατομμύριο, χρησιμοποιήστε, στείλτε 999.000 κλπ. Μη λέτε ότι μεταφέρεται ε, μάλλον εμπορεύματα από λιμάνι αν η εταιρεία σας δεν εδρεύει κοντά σε λιμάνι. Ε, έδιναν σαφείς οδηγίες για να αποφευθεί ο εντοπισμός του ξεπλήματος χρήματος. Το 2010 ξεκινήσαμε το έργο μας. Και τι είδαμε. Ότι το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το 2010 εργαζόμενοι σε άλλα προγράμματα μαζί με μια ομάδα διαφόρων ερευνητικών ε, ε, δημοσιογράφων, ερευνητών κλπ. Είχαμε αναμειχθεί και στις έρευνες που γινόταν για το έγγραφα του Παναμά, Λουξ Λίξ κλπ. Και τι, βρήκαμε τελικά το ρωσικό πλυντήριο όπως το ονόμασα. Το σύστημα της Μολδαβίας, το δικαστικό και τραπεζικό, χρησιμοποιεί το για ε, επιχειρήσεις ξεπλήματος χρήματος μεγάλης κλίμακας. 20,8 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια εστέλνοντο από τη Ρωσία και κάποιες τράπεζες που εμπλέκονται ε, συνδεόταν και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν 19 τράπεζες στη Ρωσία μία τράπεζα στη Μολδαβία και όλα τα χρήματα πηγαίναν στην Trust Κομμέρσα Μπάνκα, Ρίγα, Λετωνία και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένε Πολιτείε και σε άλλες χώρες. Το ρωσικό πλυντήριο στο σημείο υποδοχής ε, συμπεριλάμβανε πάνω από 5.000 εταιρείε, 732 τράπεζες σε 96 χώρες. Μιλάμε για όλο τον κόσμο, με άλλα λόγια. Τεράστιο το μέγεθος. Και αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν το εξετάσαμε ήταν το εξή όλα ξεκινούσαν από μια τράπεζα στη Δημοκρατία της Μολδαβία. Δύο Δύο προσεγγίσεις ακολουθείς όταν βλέπεις τέτοιες επιχειρήσεις ξεπλήματος χρήματος. Και είχαμε πάνω από 60.000 συναλλαγές. Πολύ δύσκολο να παρακολουθηθούν αυτέ. Δεν νομίζω ότι καμιά μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή κάποιο τμήμα συμμόρφωση σε οποιαδήποτε μεγάλη τράπεζα θα μπορούσε να επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία και να εξετάσει 60.000 ύποπτε συναλλαγέ. Αλλά μπορεί να το αντιμετωπίσει κανεί διαφορετικά ένα σημείο προέλευσης. Και αυτό είναι το πρόβλημα το παρόν σύστημα. Και γι' αυτό αποτυγχάνει. Έχουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Να γνωρίζουμε τον πελάτη μας κλπ. Και τον πελάτη του πελάτη. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι διευθύνς των τραπεζών που χρησιμοποιούνται όμως για να σταθούν, σταλούν τα εμβάσματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα. Ποιος είναι ιδιοκτήτης της τράπεζας στη Μολδαβία που έδινε τη δυνατότητα να αποσταλούν 20,8 δις ε, αμερικανικά δολάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα και σε άλλες χώρες μέσω εμβασμάτων. Αν δείτε την ιδιοκτησία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της τράπεζας, βλέπετε ότι είναι εταιρείε υπεράκτης, οι περισσότερες βρετανικές, SLP και LP, χωρίς να έχουν πραγματικούς δικαιούχους ιδιοκτήτες. Αν δείτε τους ανθρώπους, βλέπετε ότι οι ιδιοκτήτες, οι επίσημοι που αναφέρονται, στα επίσημα στοιχεία με τις καταχωρημένες εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεσολαβητές. Ε, αν δείτε τους δικαιούχους ιδιοκτήτες που παρουσιάζονται ότι είναι ιδιοκτήτες τραπεζικών λογαριασμών είναι οι ίδιες, οι ίδιοι φορείς. Είναι εύκολο να εντοπιστούν. Μερικά κλικαρίσματα τους ανακαλύπτεις. Δεν χρειάζεται να εξετάσεις 60.000 συναλλαγές για να καταλάβεις ότι κάτι τρέχει. Από τη στιγμή όμως που δεν γνωρίζεις ποιος είναι ιδιοκτήτης των τραπεζών που στέλνουν τα εμβάσματα και αυτό ισχύει με πολλές τράπεζες. Τώρα μιλάω για το ρωσικό πλυντήριο, τα 20 δις. Αλλά στη Μολδαβία υπήρχαν τέσσερις άλλες τράπεζες, από τις οποίες ε, ε, ε, έκλεψαν ένα δις οι εγκληματίες που έφυγαν από την οικονομία της Μολδαβίας. Υπάρχουν πολλές άλλες περιστάσεις, τις οποίες γινόταν ξέπλυμα χρήματο σε πολύ μεγάλη κλίμακα και είναι πολύ εύκολο να το πιστεί. Δεν χρειάζεται να εξετάσει τι συναλλαγές. πρέπει να προσπαθήσεις να διαπιστώσει τι γίνεται με την τράπεζα, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε τη τράπεζα. Οπότε τώρα έχουμε ερχόμαστε μεγάλε τράπεζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα χρήματα στο ρωσικό πλυντήριο ε, τα επεξεργάστηκε η Τρόστα Κομέσκ Μπάνκα που έκλεισε πέρσι την Άνοιξη μετά την υποβολή των εκθέσεών μας. Η Privat Bank επίσης είχε αναμειχθεί και η Danske Bank πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια χειρίστηκε στο όλο σύστημα. Η Deutsche ε, Bank επίση, ξέπλυνε πολύ χρήμα. Και όταν μιλήσαμε με την Deutsche Bank μα είπαν κοιτάξτε ήταν δυνατόν διότι τα χρήματα εστάλησαν μέχρι το τέλο 2014. Ε, ήταν δυνατόν πριν, διότι δεν είχαμε αρκετού υπεύθυνου για τη συμμόρφωση. Προσλάβαμε άλλα χίλια άτομα για να κάνουν αυτό να εξετάσουν τη συμμόρφωση. Αυτό δεν αρκεί κατά την άποψή μου. Ο κ. Κωνσταντσο έχει δίκιο. Πράγματι, χρειάζεται η χρήση τεχνολογίας σε αυτό το επίπεδο για να μπορούμε να εντοπίζουμε τέτοια σχήματα συναλλαγών. Είδα ένα σχήμα συναλλαγών, μορφή συναλλαγών, ότι ερευνούσαμε ξανά και ξανά το ίδιο. Και αυτά τα σχήματα και οι μέθοδοι εντοπίζονται εύκολα μέσω λογισμικού. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε τώρα στο πρόγραμμά μας. Ε, ε αναπτύσσουμε ένα σύστημα αναφοράς σχημάτων απατών. Είναι λογισμικό που μπορεί να εντοπίζει ύποπτε συναλλαγέ που μπορεί να προέρχονται από διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο και λοιπέ άλλε τέτοιε δραστηριότητε. Υπάρχει, πρέπει, να, πρέπει να δράσουν οι μεγάλες τράπεζες, πρέπει να γίνουν έλεγχοι με τις μεγάλες τράπεζες, με τις τράπεζες που έχουν κάποιους αντίστοιχους λογαριασμούς σε αυτές τις μεγάλες. Είναι εύκολο να γίνει. Η Deutsche Bank, Raiffeisen Danske, δεν, έχουν δεν υπάρχουν τόσο, τόσοι πολλοί αντίστοιχοι τραπεζικοί λογαριασμοί άλλε τράπεζες στον κόσμο. Είναι κάποιες χιλιάδες. Αυτό είναι εφικτό. Χωρίς 10.000 ανθρώπους που θα το επεξεργάζονται και πολλού πόρου. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπούρκαντς. Can start with the introductory statement. Yes, please. κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο. Uh, I am head of Latvian Financial Intelligence Unit, uh, which uh, name is uh, Office for Prevention of Laundering Procedure. Είμαι αρμόδιος για τα θέματα αυτά στη μονάδα των χρηματοϋποστατικών πληροφοριών της Λετωνίας. Το 1998 αρχίσαμε, ήμασταν μια διοικητική δομή είχαμε την ε, τη λειτουργία μας υπό την επίβλεψη του εισαγγελέα. Από το 2005 έχουμε ένα ρόλο συντονιστικό θα ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συντονίζει ο Πρωθυπουργό. και από το 2005 έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση αυτών των ε, τύπων των σχημάτων ε, ξεπλήματος χρήματος. Ε, σε διάφορες συναλλαγές επαναλαμβάνονται αυτά. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η δέσμευση των χρημάτων και η τρίτη η δρομολόγηση της έρευνας. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στι εξή στατιστικές, την τελευταία τριετία, τρισήμιση χρόνια μάλιστα. Χίλια εμβάσματα για το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού έχουν εκδοθεί για ένα συνολικό ποσό πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ σε διαφόρους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και φυσικά πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Από ξένους συναδέλφους επίσης παίρνουμε πληροφορίες και όπως δείχνουν οι στατιστικές το 2016 είχαμε ε, 34 μέρες ε, ε, προθεσμία για να λάβουμε απάντηση. απαντάμε τώρα πολύ πιο γρήγορα και συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους συναδέλφους. Τι γίνεται με τις παγωμένες ε, αυτές καταθέσεις στη Λετωνία. Το 2016 ελήφθησαν 17 αποφάσεις για πάγωμα ε, σε περιπτώσεις ποινικών διώξεων και το συνολικό ποσό ήταν 59,5 εκατομμύρια ευρώ ε, που είχαν κατασκευθεί, καθώς επίσης και αυτοκίνητα. 46 εκατομμύρια ευρώ από το ποσό αυτό ε, κατασχέθηκαν προς όφελος του κρατικού προεπολογισμού. Ωστόσο η καταπολέμηση του ξεπλήματος δεν είναι το μόνο που κάνουμε ούτε τελειώνει εδώ. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε την τέταρτη οδηγία και την προσαρμογή στο σύστημα αναφορών ε, των χρηματοπιστωτικών ε, ε, πληροφοριών για να γίνει το σύστημά μας πιο αποτελεσματικό. Αυτά ήταν τα σύντομα σχόλια που σας ανέγνωσα σχετικά με τη δράση και τη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Thank you so much. So now Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε το λόγο στους δύο συνεισηγητές πρώτα. yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Κάποιοι από εμά γνωρίζουμε αρκετά καλά την υπόθεση του ρωσικού πλυντηρίου. Εξακολουθεί όμως να είναι συγκλονιστικό το ποσό των χρημάτων και το πώς μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει με τη συμμετοχή τόσων κρατών μελών και της Μολδαβίας βέβαια στον κύριο Ράντου, θα ήθελα να απευθύνω την ερώτηση. Εσείς πώς βλέπετε αυτήν την κακοδιαχείριση από πλευράς των αρχών. Βλέπετε να υπάρχει κάτι τέτοιο στην υπόθεση αυτή και τα κράτη-μέλη που ανήκουν σε αυτή την εξίσωση. Στον κύριο Μπούλκανς. Το σκάνδαλο αυτό, ε, στο σκάνδαλο αυτό εμπλέκονται πολλά κράτη-μέλη ε, και η Δανία, πολλά εκατομμύρια πέρασαν από τις δύο τράπεζες της Δανίας. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο και στη Λετωνία. Πώς χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή, πώς ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι τράπεζές σας. Και τι συνέβη και εντοπίσατε εσείς το πρόβλημα νωρίτερα. Επίσης, μιλήσατε για τις ε, ποινικέ διώξεις. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της ε, μονάδας σας. Ε, βλέπετε όμως επαρκείς ποινικέ διώξεις και η συνεργασία της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Λιτωνίας με άλλες μονάδες άλλων κρατών μελών πώς προχωράει. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, κύριε Κόφωτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ρωσικό πλυντήριο δείχνει ακριβώς την έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα σε αρχές επιβολής του νόμου, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών κλπ. Αποκαλύψαμε το σκάνδαλο το 2014. Πέρσι, αρχές επιβολής του νόμου σε δύο χώρες ήρθαν και μας είπαν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τι έρευνε μα λόγω της έλλειψης συνεργασίας διασυνοριακά και ιδιαίτερα επειδή η Ρωσία δεν έδινε πληροφορίες. Η Ρωσία, το FSP, ζήτησε πολλές πληροφορίες, δεν μας έδωσε όμως ποτέ πληροφορίες. Μας έδωσαν λοιπόν ε, τα δεδομένα, μας ε, έδωσαν στοιχεία για τις ε, συναλλαγές και έτσι τελικά συνεργαστήκαμε με την Süddeutsche Zeitung, με την Guardian και με άλλες εφημερίδες και δείξαμε πού πήγαν τα χρήματα από το ρώσικο πλυντήριο. Η προσέγγιση ήταν να εξετάζουμε τις συναλλαγές. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι οι εγκληματίες αυτοί είναι πολύ δημιουργικοί, έχουν πολύ περισσότερη εμπειρία από κάποιον υπάλληλο μιας υπηρεσίας σε μια χώρα, διότι και διασυνοριακά έχουν πολύ εμπειρία, ε, έχουν πολύ περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους, έχουν συμβούλους, έχουν πολύ υποστήριξη για να δημιουργήσουν ε, αυτά τα προγράμματα. Το να εξετάζουμε λοιπόν τις ύποπτες συναλλαγές μάλλον μα μπερδεύει. Πιο εύκολο είναι να κοιτάξουμε τι Τράπεζε, διότι αν έχει κανεί πρόσβαση στι Τράπεζε που αποδείχτηκε ότι βοήθησαν ε, σε μεγάλη κλίμακα την ε, το, το ξέπλυμα χρήματο, ε, την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων. Αυτό θα μα βοηθήσει να πιάσουμε του εγκληματίε. Κύριε Μπούρκαν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, φυσικά. Τρει ερωτήσει θέθηκαν και θα τι απαντήσω μία προ μία. Καταρχάς, ε, πώς συνέβησαν όλα αυτά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το ρωσικό πλυντήριο πραγματοποιήθηκε από το 2011 μέχρι τον Οκτώβριο του 2014. Και βέβαια δεν μπορώ να σας ε, δώσω πληροφορίες ε, σχετικά με τους δημοσιογράφους, αλλά ήδη στις 17 Μαΐου του 2012 λάβαμε την πρώτη αναφορά σχετικά με ύποπτη συναλλαγή από τράπεζα. Δεν μου επιτρέπετε να σας αποκαλύψω για ποια τράπεζα πρόκειται, αλλά είδαμε αυτήν την αναφορά, η οποία ήταν πολύ καλή και μετά από λίγες μέρες ετοιμάσαμε έκθεση πρωτοβουλίας προς την Μολδαβία και τους είπαμε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Σας παρακαλώ, κάντε αμέσως κάτι. Ε, αλλά σιωπή. Μετά από ένα χρόνο περίπου στείλαμε δεύτερη αναφορά διότι είχαμε πληροφορίες από την τράπεζα, βλέπαμε τις συναλλαγές. Και πιστέψαμε ότι είναι θέμα νομικής βάσης. Οι δικαστές στην Μολδαβία είχαν ε, εκδώσει αποφάσεις δικαστηρίων και η βάση για αυτές τις συναλλαγές ήταν ακριβώς αυτές οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Ξεκίνησαν λοιπόν οι προκαταρκτικές έρευνες και είμαστε πολύ περήφανοι διότι πιστεύουμε ότι ήμασταν οι πρώτοι που διαπιστώσαμε ότι κάτι πάει στραβά ενώ όλοι οι συναδελφοί μας ε, άργησαν. Όσον αφορά τις ποινικέ διώξεις, θα ήθελα να πω ότι στη Λετωνία έχουμε αρκετές τέτοιες ποινικέ υποθέσεις. Φυσικά αυτές δεν είναι αρμοδιότητα της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αλλά η αποτελεσματικότητα των ε, ερευνών είναι δική μας δουλειά και η συνέχιση και οι εργασίες οι δικές μας συνεχίζονται και εργαζόμαστε σκληρά. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι τράπεζές μας εποπτεύονται από την Επιτροπή Τραπεζών και Κεφαλαιαγορών και η Επιτροπή αυτή έκανε τις δικές της έρευνες και όπως διαπίστωσαν και οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεών τους, υπήρχαν κενά στο σύστημα εσωτερικών ελέγχων. Διαπιστώσαμε λοιπόν παρατυπίες, ε, νομιμοποίηση εσόδων από παράγοντε δραστηριότητες και κενά στους εσωτερικούς ελέγχους. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν ανακάλεσε την άδεια της σχετικής τράπεζας η οποία δεν λειτουργεί πια από τον περσινό Μάρτιο. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, τη συνεργασία με άλλες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Αναφέρθηκα ήδη σε αυτό. Όταν λαμβάνουμε αίτημα για πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Ε, έχουμε εμπειρίες στον τομέα αυτών. Ήδη το 2012 ή το 2013 ήμασταν σε θέση να παγώσουμε κάποιους λογαριασμούς. με βάση τα στοιχεία που είχαμε ήδη τότε. Όσον αφορά όμως τη γενική συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, από το 1999 ε, συμμετέχουμε στην ε, ε, διεθνή οργάνωση και υπάρχει και το δίκτυο των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Θα ήθελα όμως ταυτόχρονα να αναφέρω ότι ο σημαντικότερος εταίρος μας είναι η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Μολδαβίας. Λαμβάνουμε πολλά αιτήματα και στέλνουμε μέσα σε 12 μέρες απαντήσεις. Αυτή λοιπόν ήταν η σύντομη μου απάντηση στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πίτερ Γέζεκ έχει το λόγο, ο συνεισηγητής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν και τις επιτυχείς εργασίες σας. Όπως είπατε, ακολουθείτε το χρήμα. Έχω ερώτηση σχετικά με αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με την προσέγγιση σας, τα περισσότερα χρήματα από πήγανε προς την Κίνα, το Χονγκ Κόνγκ κλπ. από το ρωσικό πλυντήριο και μικρές χώρες. Και όχι στη ΣΥΠΑ, για ποιο λόγο. Για τον κύριο Μπούλκανς, παρόμοια ερώτηση. Η Λετωνία δεν ήταν χώρα αποδέκτης των χρημάτων από το ρωσικό πλυντήριο. Γιατί? Διότι το ανακαλύψατε πιο νωρίς από τους άλλους. Το κόλπο αυτό. Ορίστε. Απάντηση. Πράγματι, βλέποντας τις ροές του χρήματος, είπα πήραν πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι άλλες χώρες. Αυτό διότι είπα είναι καλύτερες στον εντοπισμό ξεπλήματος χρήματος και γίνεται κατάσχεση χρημάτων. Μία από τις υποθέσεις που εκθέσαμε το 2010 ήταν η υπόθεση Μαγνίσκι, Μεγάλη υπόθεση σε όλη την Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ. Και τον περασμένο μήνα μόλις η εισαγγελία στη Νέα Υόρκη ήρθε συνεννόηση με την ομάδα που έκανε ε, αυτό το ξέπλυμα και κατήσχεσε 5,9 ε, δισεκατομμύρια δολάρια. Κυνηγάει το χρήμα η Αμερική. Δεν θέλω να ξεχωρίσω ότι η Λετωνία δεν είναι μόνο λετωνικές τράπεζες και άλλες χώρες παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες όσον αφορά το τραπεζικό απόρριτο. Η Λιθουανία είναι το ίδιο, η Εστονία, διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματο. Υπάρχουν πολλά πλυντήρια. Εδώ μιλάμε για το ρωσικό πλυντήριο. Υπάρχουν πολλά άλλα πλυντήρια. Στην Ουκρανία ε, ε λέγονται προσάτσκι. Είναι για ποσά περίπου ένα δισεκατομμύριο ε, δολάρια Αμερική. Υπάρχουν πάρα πολλά πλυντήρια. Άρα η γενική εικόνα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που παρουσίασα εδώ, 20 δισεκατομμύρια. Άλλοι μιλάνε για 80 δι την ίδια περίοδο. Όταν λέω άνθρωποι και κάποιοι Αναφέρομαι στις αρχές ε, επιβολής του νόμου στη Μολδαβία. Ε, πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αν δείτε τι γίνεται με τη διευθυνσία των τραπεζών, όπως σας έλεγα, εντοπίζονται προβλήματα. Αν δείτε τα αρχεία των ελβετικών τραπεζών, των λετωνικών τραπεζών, βλέπετε ότι υπάρχει κάποια ε, διάταξη να μην έχουν υπηκότητα αμερικανικοί πελάτες. Άρα ερχόμαστε τώρα στο θέμα ότι οι ΗΠΑ δεν δέχονται πολλά χρήματα. Πάνε χρήματα στις ΕΠΑ, αλλά πολύ λιγότερα. Σε κάποιε περιπτώσεις οι αμερικανικές τράπεζες αρνήθηκαν ε, συναλλαγές. Ο κύριος Μπούλκανς, θέλετε να απαντήσετε. Εγώ επισκέφθηκα τη Μολδαβία και ήρθαν και εδώ συνάδελφοι στη Ρήγα συζητήσαμε την κατάσταση. Γιατί έρχονται στη Λετωνία τα χρήματα και όχι σε άλλες χώρες. Και γιατί προτιμούν τη Λετωνία οι, οι Δεν υπάρχει κάποιος πολύ σημαντικός λόγος γι' αυτό. Είμαστε σαν γέφυρα μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών ίσως. Ίσως γιατί κατανοούμε τα ρωσικά έχουμε κοινή ιστορία λοιπά με τους Ρώσους. Αυτά είναι τα δικά μας συμπεράσματα. Χρειάζεται επιστημονική έρευνα κανονικά. Να ρωτήσουμε τις εγκληματίες γιατί προτιμάτε αυτές τις χώρες και όχι άλλες. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λίγοι. λόγοι, συγγνώμη. Για να καταπολεμήσουμε επιτυχία το ξέπλυμα χρήματος χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ καλό νομικό πλαίσιο για να παγώνουμε χρήματα για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο και να μπορούμε να συνεργαστούμε με συναδέλφους. Αν εκδίδονται χίλιες εντολές για πάγωμα ε, στοιχείων ενεργητικού, ε, παγώνουν τα ποσά μόνο για μία, δύο, τρεις μέρες. Είναι πολύ δύσκολη συνεργασία και τους καλούμε. Αν έχετε πληροφορίες, ζητήστε από μας να παγώσουμε τους λογαριασμούς. Αλλά τα... αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Κύριε Μπούλκας, Ο κύριος Ντομπρόφσκης, που είναι τώρα επίτροπος ε, Λετωνός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ήταν τότε πρωθυπουργός στη Λετωνία όταν συνέβησαν όλα αυτά και ίσως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Αλλά όπως είπε ο κύριος Ραντού, δεν είναι μόνο η Λετωνία, είναι και πολλές άλλες χώρες. Το λόγο έχει ο κύριος Ρωσάτη, τους Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να αναφερθώ στις περιπτώσεις που εσείς έχετε καταγράψει ε, στη Λετωνία και άλλο κύριε Ράντου. Και πρόσφατα ανέκυψε και ένα θέμα με μια τράπεζα από τη Σλοβενία. Ένας Ιρανός έστειλε ένα έμβασμα ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα εναντίον του και η τράπεζα το σπασε αυτό το δισεκατομμύριο και το έστειλε σε 400 λογαριασμού παγκοσμίω. η Σλοβενική. Το έχετε ακούσει αυτό, ε, έχει απασχολήσει την Επιτροπή μας και το ψάχνουμε. Αυτό είναι ο τύπος συναλλαγών στον οποίο αναφερθήκατε, το σχήμα, το συνηθισμένο. Δεύτερη ερώτηση επειδή εστιάσατε στις τράπεζες, αυτό προτείνετε, στην προσέγγισή σας. Έχουμε διάφορες οδηγίες για το ξέπλυμα, 2, 3, 4. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν μια σειρά από στοιχεία. Μας είπατε ότι υπήρξαν 60.000 ύποπτες συναλλαγές σε κάποια περίπτωση. Αυτές δεν τις ανέφεραν την ίδια μέρα, ούτε τον ίδιο μήνα. Ε, και αν αυτό ε, εμποδίζει τις μονάδες να το, τις, ε, ψάξουν τις υποθέσεις. Οι τράπεζες κάνουν τη δουλειά τους, τις αναφέρουν σωστά αυτές τις περιπτώσεις, τις ε, καταγγέλουν. Και ε, αν έχουμε πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα με την κείμενη νομοθεσία που είναι γεμάτη παραθυράκια και είναι σκέτη γραβιέρα και δεν μπορεί να εντοπίσει ε, ύποπτες πρακτικές συναλλαγές ή απλώς κάποια παράνομη συμπεριφορά. Αυτό είναι ότι δεν τα βρίσκουμε ή ότι δεν τα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη τα όσα ισχύουν. Ε, είπατε ε, ότι κάποια κράτη-μέλη είναι πιο δραστήρια ή ακούγονται περισσότερο ε, για το ξέπλυμα, ενώ κάποια άλλα δεν είναι τόσο πολύ στο προσκήνιο. Θα λέγατε λοιπόν με βάση τη δική σας εμπειρία ότι υπάρχουν διαφορές και ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Η νομοθεσία αυτή ή η εφαρμογή της. Να κλείσουμε και εμείς που νομοθετούμε ή να επιμείνουμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα και με μεγαλύτερο στένος και αποφασιστικότητα την νομοθεσία. This is, this is by the way the question. Αυτή φυσικά είναι ερώτηση και προς τον κύριο Πούρκανς. Κύριε Εγώ βλέπω μόνο τον τομέα που καλύπτει η δική μας μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Δεν έχω πληροφορίες σχετικά με τα όσα γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη μου όμως είναι ότι κάποιες άλλες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι μάλλον πιο αργές. Εάν λαμβάνουμε πληροφορίες εντός συγκεκριμένου χρόνου, αυτό θα μας βοηθήσει να ε, ενεργούμε και πιο γρήγορα. Μπορεί οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών να έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Ε, ή μπορεί κανείς να έχει να λαμβάνει πολλές αναφορές. Εμείς στη Λετωνία λαμβάνουμε 15 με 16 χιλιάδες αναφορές το χρόνο και αναλύουμε την κάθε μία από αυτές. Δηλαδή, περίπου χίλιες αναφορές ανα εργαζόμενο. Κάθε χρόνο, ε, ο κάθε χρόνος έχει κάτι λιγότερο από 300 εργάσιμες. Δηλαδή, τρεις αναφορές πρέπει να αναλύονται την ημέρα, το οποίο σημαίνει ότι ο χρόνος ανάλυσης είναι αρκετά σύντομος. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μας. Για παράδειγμα, φέτος, ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις μας και ε, Τελικά ε, τα αναφέραμε αυτά στο Υπουργείο Οικονομικών που λέει ότι δεν ε, θα πρέπει να, εξετάζουμε την κάθε αναφορά, πρέπει να τις χωρίζουμε σε είδη αναφορών. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο εργασίας δηλαδή και να εφιστούμε την προσοχή σε υποθέσεις μεγάλης κλίμακας. Ευχαριστώ. Κύριε Ραντού. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, δύσκολες ερωτήσεις. Δεν ε, γνωρίζω συγκεκριμένα ε, το θέμα της Σλοβενίας, αλλά υπάρχουν πολλά πλυντήρια και αυτό που πρέπει να καταλάβει κανείς είναι ότι πρόκειται για δομές ε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Tor. Το Tor είναι ένα εργαλείο στο διαδίκτυο για να κρύβει κανείς ε, τις ε, ενέργειες του στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να κάνω μια αναζήτηση, αυτή πηγαίνει μέσω ε, άλλων ε, υπολογιστών για να κρύψει τις κινήσεις μου. Το ίδιο ισχύει για το ρωσικό πλυντήριο και το σλοβένικο πλυντήριο. Δηλαδή, πολλές εγκληματικές ομάδες και πολιτικοί, συγκεντρώνουν τα χρήματά τους ε, και τα ξαναμοιράζουν εκ των υστέρων. Είναι mix and match που λέμε. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Ε, βλέπουμε λοιπόν το πλυντήριο ε, στη Ρωσία, βλέπουμε συναλλαγές στη Μολδαβία, στη Λετωνία και αλλού. Έτσι συγχωνεύονται τα χρήματα από το Βιετνάμ με τις Σιναλό, από το Μεξικό. Και ναι, είχαμε, θα ήθελα πολύ να είχαμε 60.000 αναφορές για υποπτές συναλλαγές, ε, αλλά βέβαια κάτι τέτοιο θα πλημμυρίσει οποιαδήποτε μονάδα οικονομικών πληροφοριών. Και άλλωστε το ρωσικό πλυντήριο είναι ένα μόνο. Ε, θα υπάρχουν λοιπόν ε, άπειρες συναλλαγές ύποπτες. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό. Εάν βελτιωθούν οι προσπάθειες σε επίπεδο μεμονωμένου κράτους, ποτέ δεν θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Χρειάζεται νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αυτό ακριβώς σκέφτονται οι εγκληματίες. Είναι οργανωμένοι εγκληματίες, δρούν διασυνοριακά. Για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια παιδική χαρά, διότι ε, τα κράτη-μέλη ε, περιορίζονται από τα σύνορά τους ε, ε, εξετάζουν ε, το καθένα τι συμβαίνει στο δικό του έδαφος. Πρόκειται για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που γίνεται με τρόπο που πραγματικά βλάπτει τις διάφορες χώρες. Βλέπαμε ότι ε, εξαίρεε το χρήμα από τη Μολδαβία επί χρόνια και δεν μιλώ για το 1 δισεκατομμύριο που εκλάπει από τις τράπεζες της Μολδαβίας. Αυτά τα χρήματα πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ψίχουλα στη Μολδαβία. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν προσέγγιση ανάλογη με αυτή των εγκληματιών. Δηλαδή ε, να ε, ενεργούμε σε πιο υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για ότα, ε, όσα μας είπατε και οι δύο είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ κατατοπιστικά. Ε, χρειάζεται δίκτυο για να αντιμετωπίσεις δίκτυα. Ε, μιλήσατε για αυτή την έννοια του να γνωρίζεις τον πελάτη σου. Έχετε στοιχεία για το ποιες τράπεζες πόσες συμμετέχουν σε αυτές τις πολιτικές. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ότι αυτά που ισχύουν ε, η αυτορύθμιση των τραπεζών δεν είναι ικανοποιητικά. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι για να το συνδέσω με την ερώτηση του κυρίου Ροσάτη. Ποιες αλλαγές ε, θεωρείτε απαραίτητες ε, στην πολιτική γνώριζε τον πελάτη σου, του Know Your Customer. Και ε, υπάρχει μια άλλη τραπέζα που ενέχεται στον Παναμά, η οποία έχει κάνει εξωτερική ανάθεση στο, στο Μόσεκ Φονσέκα κιόλα ε, αυτό το θέμα της διαχείρισης του πελατολογίου. Και ε, αυτό με τα δίκτυα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι για να καταπολεμήσεις ένα δίκτυο χρειάζεσαι δικό σου δίκτυο. Ε, τώρα που θα γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστω και περιορισμένα, ε, σε ποιο βαθμό μπορεί να ασχοληθεί, γιατί είναι ακόμα στα σπάργανα. Ενδεχομένω να μην καλύπτει ε, στο πεδίο αρμοδιοτήτων αυτό το τομέα. Τι θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράτο για την απάντηση. Ο κύριος Μπούρκανς. Ναι, με καλύψατε. οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν καλύπτουν το θέμα του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών. Είναι ευθύνη της ε, τρομοδίου φορέα ελέγχου των χρηματοδοτικών αγορών στη Λετωνία. Εμείς δεν είμαστε εποπτική αρχή. Προβληματιζόμαστε για την κατάσταση. Πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση πώς να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα του χρήματος με επιτυχία. Είχα προτείνει κάτι ήδη. Από τη στιγμή ε, προβλέπεται νομικά το πάγωμα των λογαριασμών και, στέλνουμε μια εντολή να παγώσουν τους λογαριασμούς, γιατί δεν μπορούμε να καλύτερα σε αυτό. Να πούμε η μονάδα δέχεται μία έκθεση από την τράπεζα. Και έχει νομική βάση να δώσει εντολή και να πει στείλτε τα χρήματα πίσω στη χώρα από εκεί που ξεκίνησε το χρήμα και κάνετε έρευνα στη χώρα Α, στη χώρα Β η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να έχει εξουσία όχι μόνο να παγώνει τα χρήματα, αλλά να στέλνει πίσω τα χρήματα στο λογαριασμό των θυμάτων. Πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Υπάρχουν συμβάσεις, οδηγίες κλπ. Υπάρχουν εμπόδια. Έξοχη πρόταση. Μετά από κάποια χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα εκδόσεως τέτοιες εντολής. Κύριε Ράντο. αν επανεξετάσουμε την όλη δομή που κρύβεται πίσω από το ρωσικό πλυντήριο, τι βλέπουμε. Τράπεζες που έπεσαν στα χέρια εγκληματιών στη Μολδαβία. Και τι έγινε. Η νομοθεσία στη Μολδαβία απαιτούσε αν είσαι ιδιοκτήτης πάνω από 5% μιας τράπεζας πρέπει να αποκαλύψεις ε, ποιος είναι ο δικαιούχος ιδιοκτήτης. Και τι έκαναν οι εγκληματίες. Είχαν το 4,9% 100 μέσω διαφόρων φορέων υπερακτίων. Εύκολο. Οι Μολδαβοί θεώρησαν ότι θα εξεγελάσουν τους εγκληματίες. Τι είπαν, επιβάλλαν ένα όριο του 1%. Τι έκαναν οι εγκληματίες, 0,9%. Το κλειδί ποιο είναι, διαφάνεια όσον αφορά τη διοκτησία των τραπεζών. Αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό ταιριάζει με τα μητρώα για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες κλπ. Του, του λεχθέντος. Οι εγκληματίε είναι πολύ δημιουργικοί. Και αν δείτε κάποιε από τι εταιρείε, στο χαρτί έχουν ιδιοκτήτε. Αλλά είναι απλώ ε, αχυράνθρωποι. Ή αυτοί που δημιουργούν τι εταιρείε είναι αυτοί που παρουσιάζονται σαν ιδιοκτήτε. Η αυτοι που δημιουργουν τι εταιρειε ειναι αυτοι που παρουσιαζονται σαν ιδιοκτητε Οι διαμεσολαβητη αν θέλετε. Είναι εύκολο να βρει ένα όνομα και να δει ότι κάποιο που είναι ιδιοκτήτη τη τράπεζα έχει άλλε 2.000 εταιρείε, άρα πού να τι χειριστεί. Η ιδιοκτησία των τραπεζών είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Σημαντικό να εντοπιστούν οι κόμβοι στα δίκτυα. Αν δούμε τι έγινε το ρωσικό πλυντήριο και μετά άλλα πλυντήρια. Πάντα υπάρχει μια χούφτα εταιριών που είναι κομβική σημασία στο σύστημα. Σαν άξονε. Στο ρωσικό πλυντήριο με τα 20 δι έχουμε να κάνουμε 12 εταιρείε. Οι περισσότερε από αυτέ είτε οι βρετανικέ ή κυπριακέ, είτε από το Delaware. Εξετάζοντα αυτέ θα έκανε τεράστια διαφορά. Μια τέτοια εταιρεία. Είναι Westburn Enterprises Limited. Βρετανική εταιρεία. Πάνω από τρία δις αμερικανικά δολάρια χειρίστηκε εντό του πλυντηρίου και σε άλλα κόλπα. Η διοκτησία ενός ενδιάμεσου ήταν αυτό. Και αυτός έδινε και τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού και τον ιδιοκτήτη της τράπεζας που παρουσιαζόταν. Αν δείτε καλύτερα τι υποδομέ, όχι τι συναλλαγέ. Δύσκολο να ακολουθήσει κανεί συναλλαγέ. Αν δει ποιο είναι ο πραγματικό ιδιοκτήτη των βασικών εταιριών και των διαφόρων ενδιάμεσων που αναμειγνύονται και αν δείτε την όλη δομή, έχουμε πέντε τέτοιου φορεί που χειρίστηκαν το όλο σύστημα τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν είναι πάνω από πέντε. Βρετανικού φορεί από τον Παναμά και με έδρα την Κύπρο και τον Delaware μια χούφτα μπορεί να ερευνηθούν. Στη ρίζα του προβλήματος που να πάμε αντί να παρακολουθήσουμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του κατακλυσμού πραγματικά των συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ο κ. Ρόμπερτ Τσίλε του ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ανάμεικτα αισθήματα διότι είμαι Από τη μια δεν αισθάνομαι και μεγάλη υπερηφάνεια. Ταυτόχρονα είναι καλό που συζητούμε το θέμα σήμερα και είναι και εδώ ο κ. Μπούρκαντς. Ο, ίδιος, ο Μπούρκαντς είπε ότι, αν, ότι η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών δημιουργήθηκε το 1998. Και θέλαμε και τότε ήμουν υπουργό οικονομικών και θέλαμε να κάνουμε τι αλλαγέ για να πλησιάσουμε κάπω τα πρότυπα τα δυτικοευρωπαϊκά σε αυτέ τι τράπεζε. Πέρασαν 20 χρόνια. Και υπάρχει και εποπτική αρχή που εξετάζει τι κεφαλαγορέ και τι τράπεζε. Δημιουργήθηκε τότε. Ερευνήσαμε το βρετανικό σύστημα εποπτείας του χρηματοδοτικού συστήματος. Το 1998 κάναμε την ερευνά. Ποιο με μπερδεύει. Αυτό περιέγραψε ο κ. Μπούρκαν, το σύστημα. Οι μονάδες ε, δεν έχουν αρκετές ε, εξουσίες. Ε, εντοπίζουν το χρήμα, παγώνουν τους οργανισμούς, δεν παστήλουν πίσω τα χρήματα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους ιδιοκτήτες τραπεζών. Και η δική μας υποπτική επιτροπή θα μπορούσε να εργαστεί με τον κύριο Μπούρκανς. Είναι μικρή χώρα η Λετωνία. όσον αφορά με τους θεσμούς που κινούνται εκεί, αλλά όχι όσον αφορά τα ποσά που ξεπλένονται. Αυτό μας ντροπιάζει. Γιατί έρχονται στη χώρα μου. Δεν είναι μόνο το θέμα, γιατί έρχονται οι Ρώσοι εδώ, δεν είναι μόνο η, γνώση των α, Ρωσικών. Αλλά έχουμε και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που είχε επηρεαστεί από τους Ρώσους. Από την παλιά εποχή. προσπαθούν ε, έχουμε το μισό των καταθέσεων που έρχονται από τρίτες χώρες φανταστείτε από ποιες χώρες ε, κατατίθενται τα χρήματα στις τράπεζες μας Και βέβαια να εξαφανιστούν πολύ γρήγορα αυτές οι καταθέσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στις τράπεζες. Έχουμε πρόβλημα συμμόρφωσης. Κάποιες από τις τράπεζές μας είχαν κάποιες αντίστοιχες τράπεζες, αμερικανικές τράπεζες για να κάνουν συναλλαγές εδώ και δέκα χρόνια. Εξαφανίστηκαν όμως αυτοί οι λογαριασμοί. Τελευταία ήταν η Deutsche Bank που είχε αναμειχθεί και τώρα έληξε και αυτό. Συνεχίζεται όμως αυτή η ιστορία. Και έρχομαι στις ερωτήσεις. Mm. Κύριε Μπούρκανς, Είπατε ένα παράδειγμα, θέλετε να μπορείτε να στείλετε χρήματα πίσω, να επιστρέψετε χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας δώσει τις εξουσίες ή μπορεί να το κάνουμε οι ίδιοι στη Λετωνία μέσω εθνικής νομοθεσίας. Δεν θα αντιβαίνει την ε, διεθνή νομοθεσία αλλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπορεί να γίνει εν μέρη και σε εθνικό επίπεδο αυτό που θέλετε ή πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να επηρεάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά και για τους δύο ερώτηση. Το βλέπετε ότι δεν θα κατανομάζεται στο μέλλον η Λετωνία σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις ε, και ανάμειξη σε επιχειρήσεις πλυντηρίων χρήματος. Λοιπόν, ο κύριος Μπούκανς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όχι μόνο μπορούμε να αλλάξουμε την εθνική μας νομοθεσία, διότι θα πρέπει να είναι δυνατή η συνεργασία με άλλες μονάδες ε, χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Καλό θα είναι να τροποποιηθεί η οδηγία, ακόμα καλύτερο θα είναι όμως να τροποποιηθούν οι συστάσεις. Θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους όλες οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτή είναι η απάντησή μου. Um, yeah, just... Κύριε Ράντου, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Η Λετωνία, όπως καταλαβαίνετε, έχει συμπεριληφθεί σε πολλές από τις εργασίες μας τα τελευταία 8 χρόνια λόγω των προβλημάτων εκεί. Βλέπω όμως ότι η Λετωνία αναλαμβάνει μέτρα κατά της ε, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Κλείνει τράπεζας, για παράδειγμα, ανακαλεί τις άδειές τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την Ουκρανία, διότι η Ουκρανία πολύ πιθανό είναι να είναι η νέα Λετωνία, Λιθουανία ή Εστονία. Υπάρχουν τράπεζες τώρα στην Ουκρανία που αναλαμβάνουν, που, ε, τις οποίες έχουν αναλάβει οι ίδιοι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε εδώ. Και μάλιστα μία από τις τράπεζες ήδη βρίσκεται στην Ουκρανία και επειδή η Ουκρανία είναι τώρα το αγαπημένο παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επιτρέψει στους οργανωμένους εγκληματίες της χώρας αυτής να συνεχίσουν τις δουλειές τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέσπο. Ερμπάν Κρέσπο, ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντάς σας, κυρίως τον κύριο Ράντο, μου έρχεται μια ερώτηση και μια παρατήρηση στο μυαλό. Εξαίρεση αυτό ή ο κανόνας. Και αυτό είναι ενισχυτικό γιατί είναι μάλλον ο κανόνας πέραν του συγκεκριμένου παραδείγματος. Και μια από τι ερωτήσεις που, για τα θέματα που μας εξέπληξαν με τα έγγραφα του Παναμά είναι ότι οι μεγάλες περιουσίες, οι μεγάλοι εγκληματίες δεν χρειαζόταν να πάνε καν ούτε στην Ελβετία ούτε στον Παναμά. Θα μπορούσαν να κατεβούν στην τράπεζα της γειτονιάς, στο πρώτο υποκατάστημα της εγωνία και με μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα να δρά ως διαμεσολαβητής και μάλιστα ως διευκολυντής για να ξεπλύνουν χρήματα ή να ε, αποφύγουν τη φορολογία, εξού και το ρωσικό πλυντήριο. Εμείς πώς θα νομοθετήσουμε σε σχέση με το ρόλο που έχουν οι τράπεζες που διευκολύνουν και το ξέπλυμα και τη φοροδιαφυγή και αποφυγή. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και στην Επιτροπή μας και στην πολιτική ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε πάρα πολύ για την τελική έκθεση. Και θέλω και στους δύο να θέσω υπόψη, ιδιαίτερα στον κύριο Ράτου, ε, το εξή και να κάνω τις εξή ερωτήσεις. Δύο. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, κατέθεσε μία πρόταση για επιβολή κυρώσεων και προστήμων στους διευκολυντές, όχι μόνο στις τράπεζες και τους λοιπούς. Αλλά επειδή είναι χαμηλό το πρόστιμο, αυτό πιάνει τόπο όταν είναι μικρές οι συναλλαγές και όχι μεγάλου βεληνικούς. Εσείς πιστεύετε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα βοηθούσε? Ε, ακόμα και για να νομιμοποιήσει τέτοια ξεπλήματα, γιατί σου λέω ο άλλος πληρώνω το πρόστιμο που είναι πενταροδοκάρες και ξεπλένω και τη συναλλαγή την ίδια. Αυτό είναι λοιπόν ε, αποτρεπτικό επιχείρημα ή χρειάζεται η φοβέρα ότι θα σου πάρω την άδεια αν συνεχίσεις και να επαναλαμβάνεις αυτές τις δραστηριότητε. Και μετά, επειδή υπάρχει και το θέμα της δέουσας επιμέλειας, γίνονται καλοί έλεγχοι εσωτερικοί από τις τράπεζες τις ίδιες. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις ότι η λεγόμενη αυτορύθμιση δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ποια άλλα μέτρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ακριβώς για να εκτελείται αυτή η ιδέουσα επιμέλεια από πλευρά των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ραντού. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε και να δούμε ποια είναι η υποδομή. Αυτοί οι διευκολυντές, εκείνοι που στείνουν τις δομές, είναι οι πυλώνες ε, του όλου συστήματος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί εκεί είναι η ισχύ του οργανωμένου εγκλήματος, ότι δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά αυτό είναι και αδυναμία. Γιατί είπατε ότι μπορείτε να πάτε στην τράπεζα της γειτονιάς εδώ, ε, στις Βρυξέλλες ε, και στη Γερμανία, είπα κατά λάθο γιατί εγώ είμαι Γερμανός από το Βερολίνο και ε, να, φτιάξετε μια δομή που συνδέεται με τον Delaware, την Εβάδα, την Κύπρο ή τον Παναμά. Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ε, δίκτυα και εκείνοι που φτιάχνουν τις εταιρείε. Η Φωσέκα είναι μια εταιρεία που έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο. Τα ίδια και στη Λετωνία και στην Εστονία. Δεν δρούν μόνο εντός των ορίων μιας χώρας, έχουν και γραφεία και συναλλαγές παντού και συνδέονται με άλλους formation agents, δηλαδή ε, ε, φορείς που ιδρύουν τέτοιες εταιρείες. Και μπορεί κάποιος να πει ότι μια εταιρεία είναι ύποπτη γιατί την έχει ιδρύσει ο τάδε ε, ατζέντης, πράκτορας εκεί. Για τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, συμφωνώ μαζί σας, τα πρόστιμα δεν είναι αποτρεπτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί όταν μιλάμε για χοντρό ξέπλυμα τι κάνουν οι εγκληματίες. Συμπεριλαμβάνουν στα έξοδα και στο κόστος και το πρόστιμο. Δηλαδή το αφαιρούν από το τελικό του κέρδος. Το κάνουν πολλές φορές. Ε, υπάρχει μια περίφημη και πολύ γνωστή περίπτωση στις ΗΠΑ και αλλού. Για τους εσωτερικούς ελέγχους των τραπεζών, τραπεζών δεν αρκούν αυτοί, διότι όπως ακούσαμε εδώ δεν έχουν αρκετό προσωπικό για να κάνουν αυτή τη βαθιά έρευνα και τον ε, έλεγχο στις επιθεωρήσεις των τραπεζών, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλο έλεγχο αυτό. Και δεύτερον, πολλές τράπεζες υποδίονται ότι το κάνουν αυτό. Έχουν κάποιες τράπεζες δεδομένων για τις ε, διάφορες ύποπτες ε, συναλλαγές και δεν ψάχνουν τον πραγματικό δικαιούχο για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και κάτι τέτοιο υποτίθεται ότι ψάχνουν, αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Ο κύριος Μπούρκανς. Yes, Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Το θέμα είναι οι τράπεζες. Μπορούμε να τους τιμωρήσουμε, τιμωρήσουμε τις τράπεζες αν δεν έχουν καλό εσωτερικό έλεγχο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που οργανώνουν αυτά τα κόλπα κατανοούν άριστα τις αρμοδιότητες που έχουν οι δυνάμεις και οι θεσμοί του νόμου. Πρέπει να στέλνουμε επιστολές για να λάβουμε μέτρα. Έχουμε σύνορα. Αυτοί δεν έχουν σύνορα. Στέλνουν τα χρήματα από τράπεζα σε τράπεζα. Και η τράπεζα βλέπει ένα κομμάτι. Εισερχόμενη και εξερχόμενη συναλλαγή. Και αν αλλάζει αμέσως χώρα το χρήμα μετά, υπάρχει άλλη τράπεζα που βλέπει την ίδια εικόνα. Πιστεύω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορά τις τράπεζες πρέπει να αυξηθεί, να διευρυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, να φαίνεται η εικόνα του δικτύου. Για την ώρα πολλές ε, Μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών αναμειγνύονται, αλλά δεν υπάρχει μία μονάδα που είναι αρμόδια για τη σε όλου του συστήματος. Ίσως χρειάζεται μία μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύστημα του πλυντηρίου καλύπτει πολλές χώρε. 96 χώρε. Έχουμε σε επίπεδο παγκόσμιο ε, ε, μονάδε σηματοοικονομικών πληρωμών. Χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σύντομα, ο κύριος Ορμπάν Κρέσπο. Ε, και η αφαίρεση της άδεια που σας ρώτησα, πιστεύετε ότι είναι αποτρεπτικό μέτρο? Θα ήταν καλό αυτό να το υποβάλουμε εμείς σύσταση σε περίπτωση που υποτροπιάζουν οι τράπεζες να τις κλείνουμε. Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οι τράπεζες να έχουν αυτό να επικρέμεται. Ο μόνος τρόπος για να συμμορφωθούν. I agree. Fully agree. Συμφωνώ απόλυτα, λέει ο κ. Κυρία Άντια Οτάλα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλο το απόγευμα ακούμε για τα κενά που υπάρχουν ε, στις ε, μονάδες συμμετοοικονομικών πληροφοριών. Κανείς δεν ανέφερε το Eurojust. Ο κ. Μπούρκανς γνωρίζει αν υπάρχει συμμετοχή του Eurojust, αν βοηθά στην διερεύνηση των υποθέσεων. Πήγα στο αρχηγείο του Eurojust μια φορά και ήθελαν πολλοί να μπορούν να συμμετάσχουν. Αν του είπε το μια αίτηση, είτε από κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ή ε, κράτο ε, που έχει ε, συμφωνία συνεργασία με το Eurojust, όπω είναι η Μολδαβία. Αυτή είναι η ερώτηση του κύριου Μπούρκαντ. Δύο σύντομε ερωτήσει στον κύριο Ράντο εξηγήσατε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών. Είπατε ότι είναι πανεύκολο να βρει κανείς τους αντίστοιχους κατόχων λογαριασμών. Χαίρομαι πολύ αν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπορείτε να το εξηγήσετε γιατί είναι τόσο εύκολο το ζήτημα και γιατί είναι τόσο εύκολο. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στην αρχική σας ανακάλυψη από την νεοζηλανδική εταιρεία στο λογαριασμό στην Λετωνία και ανήκανε τα χρήματα σε Ρώσους εγκληματίες και κάποια ανήκανε στο, στην περίπτωση Μαγνίσκη. Πρόσφατα στο CNN και σε άλλα ΜΜΕ αμερικανικά αναφέρθηκε ότι κάποια τα χρήματα Μαγνίσκη όπως αποκαλούνται εντοπίστηκαν σε κάποια προγράμματα για χημικά όπλα στη Συρία. Ξέρετε κάτι? μπορεί να βρεθεί αυτή η σχέση με κάποιο να διαπιστωθεί ότι πράγματι υφίσταται με αξιόπιστο τρόπο είναι απλώ μια υπόθεση, μια θεωρία. Κύριε Μπούρκαν, σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη είπα ότι από το 1998 είμαστε μέλη της ομάδας Egmont όπου συμμετέχουν πάνω από 50 μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ανταλλάσσουμε πληροφορίες μεταξύ μας. Αυτό είναι σημαντικό δίκτυο για μας. Φυσικά, ε, εάν είναι απαραίτητο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το FIUNet ή να ανταλλάξουμε πληροφορίες μέσω της Interpol, της Europol ε, ή ακόμα και να υποβάλουμε αίτημα στην Eurojust. Αλλά το βασικό δίκτυο για μας είναι η ομάδα ΕΚΜΟΝ, το που συμμετέχουν 150 μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ναι, η πρώτη μου ερώτηση. Ε, μάλλον η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Τράπεζες, ε, όχι. Οι τράπεζες ε, πρέπει να το εγκρίνουν οι μικρές τράπεζες, δηλαδή πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό σε μεγάλη τράπεζα για να έχουν πρόσβαση στο διεθνές ε, χρηματοοικονομικό σύστημα, για να μπορούν να μεταφέρουν χρήματα. εμείς πώς εντοπίζουμε τις αντίστοιχε τράπεζε, Οι περισσότερε από αυτές είναι δημόσιες, διότι οι μικρές τράπεζες ε, ε, διαφημίζουν στις ε, ιστοσελίδες του ότι εμείς έχουμε επαφή με την Τράπεζα τη Νέα Υόρκης και με άλλες μεγάλες τράπεζες. Από δικαστικές υποθέσεις και από διαρροές πληροφοριών καταφέραμε να εντοπίσουμε τους κωδικούς SWIFT και τους κωδικούς των εμβασμάτων. Το πολύπλοκο στα πλυντήρια είναι ότι έχουν αναμειχθεί χρήματα από διάφορες πηγές. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό το ε, πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας να χρηματοδοτήθηκε από εδώ, διότι ε, στη Νέα Ζηλανδία είδαμε χρήματα από τη Συναλό, ε, ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ ναρκωτικών της, του Μεξικού και είδαμε ότι ένας Βιετναμέζος ε, ε, μας εξηγούσε πώς μετέφερε χρήματα, διότι ήταν στη φυλακή στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να δει κανεί τι μπαίνει και τι βγαίνει, αλλά είναι πολύ πιθανό, ναι, πράγματι να ισχύει αυτό, ότι ε, να χρηματοδοτήθηκε ε, με τέτοιο χρήμα. Είδαμε και πολλά χρήματα από το Ιράν ε, στις έρευνες αυτές. Η κυρία Γκόμες, ναι, σειρά μου τώρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια πιθανότατα να μην αρκεί για τους μετόχους των τραπεζών στη χώρα μου, στην Πορτογαλία. Ε, ούτε όταν ήμασταν υπό την εποπτεία της Τρόικας γίνονταν ε, έρευνες ε, σχετικά με τους μετόχους ε, και γίνανε αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να γίνουν έρευνες, αλλά δεν έχει κλείσει το θέμα. Όσον αφορά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και την απόσυρση της άδεια των τραπεζών και όχι μόνο των τραπεζών αλλά και διαμεσολαβητών όπως είναι οι δικηγόροι. Η ερώτησή μου είναι Πώς βλέπετε το σύστημα, το αγοράζει κανείς την άδεια παραμονής του στην ε, Ευρώπη. Ε, κατόπιν μπορεί να υποφεληθεί κανείς από τα κέρδη του πλυντηρίου ή είναι αυτό τμήμα του, του Νομίζω ότι τα προγράμματα με τις χρυσές θεωρήσεις επιτρέπουν σε χρήματα από το πλυντήριο να εισέλθουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς ε, δεν ε, θέτει κανείς πολλές ερωτήσεις στη στιγμή που μπουν τα χρήματα στη χώρα. Εκδίδεται η θεώρηση και συνεχίζουμε κανονικά. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά έχει πολύ σημαντικές αντικές επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Κύριε Μπούρκανς, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Για παράδειγμα, η δική σας μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, μπορεί να εξετάσει τι γίνεται με το δικό σας πρόγραμμα επενδυτών. Ναι, το εξετάζουμε το θέμα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι έχουμε στείλει αρκετές υποθέσεις στον εισαγγελέα, αλλά ο αριθμός αυτών των υποθέσεων είναι πολύ περιορισμένος. Σε πολλές περιπτώσεις, ε, άλλωστε, είναι καθαρό το χρήμα, αλλά μαζί με την αστυνομία εξετάζουμε καθημερινά τις υποθέσεις αυτές και με τη βοήθεια λογισμικού καταφέρνουμε να βρούμε τα ε, τα έσοδα από έγκλημα. Ο κύριος Νούνο Μέλος στη διαδικασία ΚΑΣΔΙΑΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούγοντας τη δική σας ερώτηση και την απάντηση, μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ερώτηση. Μιλάμε με βεβαιότητα, αλλά καμιά φορά αντιμετωπίζουμε περιστάσεις που είναι διαφορετικές. Το θέμα του προγράμματος αυτού των θεωρήσεων ήταν ένα σχήμα για ξέπλυμα χρήματος. Στην Πορτογαλία το πορτογαλικό δίκαιο επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις ένα πάγωμα όταν δημιουργούνται εταιρείε και δημιουργούνται θέσεις απασχόλης δίνεται αυτή η θεώρηση δεν είναι μόνο για ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι εποφελές και για τη χώρα. Δημιουργούνται εταιρείε στη χώρα μας, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, άρα ε, είναι κάτι εποφελές. Δεν νομίζω ότι καλύφθη αυτό από την απάντησή σας. Θα μου πείτε ότι ίσως υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα και δεν υπάρχει βεβαιότητα. Δεν υπάρχουν βεβαιότητε. Η πραγματικότητα ποικίλει. Δεν θεσπίζω εγώ του κανόνε. Ερευνώ και αποκαλύπτω αυτά τα τεχνάσματα, τα εγκληματικά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πρώτα η Αμερική και αποσύρισα τη Συμφωνία των Παρισίων, η Λετωνία πρώτη, Εστονία πρώτη, η Πορτογαλία πρώτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται. Αυτό είναι. Εκεί καταλήγουμε. Με τα προγράμματα της χρυσή θεώρησης της βίζας προσελκύει επενδυτές εις βάρος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ανάλογα με το τι προσφέρεις. Όπως τα βλέπετε εσείς, αν είσαι, είσαστε μια χώρα που προσελκύει τέτοια χρήματα, αυτό είναι καλό για σας, εντός συνόρων σας. Δεν λέω ότι όλα αυτά είναι βρώμικα χρήματα. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι καθαρά χρήματα. Παρά την ηθική επιχειρηματολογία αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για το οργανωμένο έγκλημα να επενδύσει. Δεν λέω ότι όλα αυτά τα χρήματα που από το οργανωμένο έγκλημα. Ο κύριος Μπόρκανς, θέλετε να προσθέσετε τίποτα? Θα ήθελα να προσθέσω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι πλυντήριο ρωσικό είτε όχι, οι δικές μας προσπάθειες εστιάζονται στο πόσο καλή είναι η συνεργασία με άλλες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Και με έχει προβληματίσει αυτό. Γιατί στην περίπτωση του ρωσικού πλυντηρίου. Γιατί δεν πήραμε καταγγελίες από τη Μολδαβία, τη Ρωσία ή από αλλού. Αλλά από τρίτες χώρες που μας είπαν ακολουθήστε το χρήμα, παγώστε τις καταθέσεις. Οι άλλοι σιωπούν. Για ποιο λόγο. Well, thank you, Ευχαριστώ κύριε Μπορχάνς. Νομίζω εδώ ολοκληρώνω τη συζήτησή μας και μπορώ να πω προφανώς ότι είναι πολύ καλό να δημιουργούνται θέσεις εργασίας στις χώρες μας. Αλλά δεν μπορούμε να καλέσουμε κάποιον από ένα ε, καρτέλ ναρκωτικό να έρθει να επενδύσει. Θέλουμε τέτοιες θέσει εργασίας που να δημιουργούν κάποιοι ναρκέμποροι ή άλλοι με το βρώμικο χρήμα. Ότι φέρτε επενδύσεις και ό,τι να είναι. Υπάρχουν και καθαρά χρήματα. Είναι ανάγκη να έρθει το βρώμικο χρήμα να επενδύει. Και να πυροδοτεί όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω θέλω να επανέλθει ο κύριος Μέλο από ό,τι βλέπω. Ένα διαδικαστικό για άλλο θέμα, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. για μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, κατανοώ αυτό που λέτε. Ε, υπάρχουν ε, εδώ ενδεχομένω πολιτικές διαφορές, ε, ανάλογα με τη σκοπιά που το βλέπει ο καθένας. Αλλά αυτό που εμένα μου φαίνεται ε, στρεβλό και διαστραμμένο είναι ότι ε, έρχεται ένας έντιμος επενδυτής να επενδύσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Και η χώρα μου δεν είναι μια περιφέρεια της Ευρώπης, είναι κυρίαρχο κράτος. Και δεν μπορούμε ε, έντιμους επιχειρηματίες να τους θεωρούμε επικεφαλής ενός καρτέλ ναρκωτικών, ας πούμε να τους συμπεριφερόμαστε σαν να ήταν τέτοιοι. Εν πάση περιπτώσει, να πω κάτι για την αποστολή στη Λισαβόνα. Να τα πω τώρα ή όταν θέλετε, Πρόεδρε, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα βιβλίο, μια, μια, μια δημοσίευση που θέλω να σχολιάσω ε, που, και απευθύνεται στους βουλευτές που θα μεταβούν στη Λισαβόνα. Το διάβασα με μεγάλη προσοχή, αλλά δυστυχώς και το έχει διαπιστώσει και ένας άλλος βουλευτής βλέπουμε κάποια άρθρα που έχει δώσει ο αριστερός συνασπισμό στον μπλόκο, της, μπλόκο Ισκέρδα, το Ισκέρδα.net, που είναι μέλη της ΓΟΕ, οι βουλευτές του. Σε αυτά τα άρθρα παραπέμπει. Βλέπω ότι σας μιλάει η βοηθό σας. Έλεγα λοιπόν ότι τα άρθρα που αναφέρονται εδώ είναι αριστερά προσκύμενα και κάποια άλλα που έχει γράψει η κυρία Αναγκόμες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά το κοινοβούλιο εδώ δεν υιοθετεί απόψεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Συνασπισμού της Αριστεράς, τον πλόκο της κέρδα της Γκουε. Εμείς έχουμε ε, μια γκάμα πολιτικών και κομματικών απόψεων υπάρχουν και άλλα άρθρα για να ενημερώσουμε τους ευρωβουλευτές που θα πάνε στην ε, Πορτογαλία. Έχει και υπηρεσίες μεταφραστικές το Κοινοβούλιο και τα Πορτογαλικά είναι επίσημη γλώσσα και μπορεί κανείς να βρει ένα οποιοδήποτε πορτογαλικό άρθρο και να το μεταφράσει στα αγγλικά. Δεν είναι επιχείρημα ότι δεν έχουμε άρθρα στα αγγλικά. Τα μεταφράζω και εγώ αν θέλετε. Λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει ε, κάποιες απόψεις κομματικές, αριστερές και δεν το θεωρώ σωστό, σαν να ήταν θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαφωνώ. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε γιατί έχει συμβεί αυτό και να ληφθεί υπόψη ότι και τα πορτογαλικά είναι επίσημη γλώσσα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι όλα στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα το διαβιβάσω αυτό στον Πρόεδρο Λάγκε. Εγώ τον αντικαθιστώ, δεν έχω καμία σχέση με τη σύνταξη αυτού του κειμένου. Υποθέτω ότι θα σα απαντήσει ο κύριος Λάγκε. Συνεχίζει στα αγγλικά η Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και οι προτάσεις που μας κάνετε ε, για την εξεταστική μας Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις 3 Ιουλίου. Με την Επίτροπο κυρία Γιούροβα και στις 10 Ιουλίου θα συνεδριάσουμε με τους Υπουργούς Οικονομικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ωράριο που θα ανακοινωθεί. Ευχαριστώ.